Ε, Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Βλέπω, βλέπω αμέσως να βάλετε τα ακουστικά. Μετά διδόμαστε και στο διαδίκτυο. Θα έχουμε τουλάχιστον 100.000 θεατές που ενδιαφέρονται να δουν τι γίνεται σήμερα στην Επιτροπή μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμα και Ισπανίος, συνάδελφος Τσέρκας Σέρκας έβαλε τα ακουστικά. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική ακρόαση δύο επιτροπών. Η μία της Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων και η άλλη είναι η, κοινωνική, η γεωργική πολιτική που θα επεξεργαστούν ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα απασχόληση για τους εργαζομένους του χώρου της γεωργίας. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι όλα πάνε καλά έχουν ε, πολλά λεφτά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια απλούστευση, υπεραπλούστευση της ε, κατάστασης. Βεβαίω και θα πρέπει να ακούσουμε θέλουμε να ακούσουμε από τους ε, γεωργούς, από τους εργαζόμενους του χώρου της γεωργίας, την, την βεβαίωση ότι οι επιδοτήσεις τους βοηθούν να παράγουν καλύτερα και πιο υγιή προϊόντα. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα με τις δύο επιτροπές μας να συναντηθούμε για να οργανώσουμε αυτή την κοινή ακρόαση. Και ο κύριος Έλγουαρθ βεβαίως είναι εδώ. Χαίρομαι που είχατε την ευκαιρία να έρθετε. Είσαστε πολύ σημαντική προσωπικότητα της Επιτροπής Γεωργίας. Βλέπω και τον κύριο, την κυρία Μαγκίνες που είναι κοντά μου πάντα καθισμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Ιρλανδή, μία χώρα, η Ιρλανδία, την οποία, για την οποία έχω μεγάλο σεβασμό, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλα κράτη. ορίζουμε. χαιρετίζουμε και τους γεωργούς της Ιρλανδίας όπως και αυτούς της Γερμανίας και όλων των άλλων κρατών. Να δούμε λοιπόν τα πρακτικά ζητήματα της δουλειά μας. Θα ήθελα να δώσω στον συνάδελφο κύριο Έλουαρτ την ευκαιρία να κάνει μια σύντομη παρέμβαση και αφού ακούσουμε και τους ειδικού μας, με μέγιστο όμως 10 λεπτά για τις ε, εισηγήσεις τους. Ξέρω ότι 10 λεπτά μπορούν να σας φανούν πολύ λίγα, αλλά να σας καθησυχάσω, οι ευρωβουλευτές πολύ συχνά έχουν μέχρι 2 λεπτά χρόνο ομιλίας, μέσα στα οποία 2 λεπτά προσπαθούν να εξηγήσουν ε, πώς γυρίζει ο κόσμος. Ενώ εσείς έχετε 10 λεπτά για να μιλήσετε μόνο για τη γεωργία και τους γεωργούς. Κύριε Έλγουαρτ, έχετε εσείς το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ με χαρά σας βλέπω εδώ όλους ε, στο σεμινάριο αυτό για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο της γεωργίας. Είχαμε προτείνει μια έκθεση πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση ευρωπαϊκού επίπεδο της ε, υγείας και ασφάλειας. Εν τω μεταξύ, 21 ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιρλανδία και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν λόγω ατυχημάτων στην εργασία στο γεωργικό τομέα, φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάθε άλλος τομέας έχει και η γεωργία του κινδύνους της. Δουλεύουμε πολλές ώρες, σκληρές ώρες, με σκληρές καιρικέ συνθήκες, με μηχανολογικά, με ηλεκτρικά, ε, τεχνικά ε, ζητήματα μπορεί να προξενήσουν ε, ασθένειες και στο αναπνευστικό Έχουμε εργασία σε απομονωμένες περιοχές, απομακρυσμένες από τον υπόλοιπο κόσμο περιοχές της εκμεταλλεύσης. Τα προβλήματα λοιπόν είναι όχι ίσως διαφορετικά, αλλά πάντως η κίνδυνη είναι πολύ πιο υψηλή και συνήθις. Κίνδυνοι που έχουν να κάνουν και με το χώρο εργασίας, αλλά και με την οικογένεια και την στέγη. Έχουμε μεγάλες, μεγάλα ποσοστά θανάτων ακόμη στους νέους και ιδιαίτερα σε παιδιά λόγω των γεωργικών ε, εργασιών. Πολύ συχνά ε, εμφανίζονται φαινόμενα παραμέλησης της υγείας, των όρων της υγείας και ασφάλειας ε, στη γεωργία που όμως έχουν τόσο μεγάλη σημασία και γι' αυτό περιμένω να έχουμε μια καλή ανταλλαγή απόψε εδώ σήμερα. Ο στόχος είναι να δώσουμε μια νέα όθηση για να προαγάγουμε την ε, ασφάλεια στην γεωργία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως είτε μαζί είτε χωριστά η κάθε επιτροπή να ε, αποφασίσουμε και την κατάρτιση εκθέσεως. Οι ομιλητές μας λοιπόν σήμερα είναι ο κύριος Πάκρη από την Υπηρεσία ε, Υγείας και Ασφάλειας της Ιρλανδίας που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό έχει εργαστεί και με, σε, πάνω σε νομοθετικές προτάσεις, κατευθυντήριες γραμμές, προγράμματα εφαρμογής. Είναι σύμβουλος στις αρμόδιες αρχές εποπτείας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι στη Μόνιμη Επιτροπή, είναι στην ΆΤΕΞ και σε άλλους φορείς που παρακολουθούν την εφαρμογή των κανόνων για την υγεία και ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης θα ακούσουμε τον κύριο Δελγάδο Κόντας από την Ισπανία, ο οποίος ε, είχε στο Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας τις αρμοδιότητες της παρακολούθησης των ε, συνθήκων υγείας και ασφαλείας και της τήρησης των όρων και την προετοιμασία ενός μη δεσμευτικού κανόνα, οδηγού καλύτερα για τα θέματα αυτά στη Γεωργία. Επίσης, έχουμε εκπροσώπους από διάφορους τομείς όπως η Διεθνής ε, Ένωση ε, Υγείας και Ασφάλειας. Έχουμε ε, δραστηριοποίηση σε θέματα υγεία και ασφάλειας στην Γεωργία και τώρα ε, θα ήθελα μετά την εισαγωγή αυτή να δώσω το λόγο στον κύριο Γκρίφιν να μας κάνει την παρουσίασή του. Παρακαλώ. Uh, thank you very much, uh, Firstly... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα. Θα αναφερθώ στο ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στον τομέα της γεωργίας, κοιτώντας κυρίως την Ιρλανδία αλλά και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μου, πάντως έχω μαζί μου και ένα φυλάδιο το οποίο μπορώ να σας δώσω, μια δημοσίευση του δικού μου του Ινστιτούτου. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι 145 γεωργικές μονάδες έχουμε στην Ιρλανδία και στο 92% αυτών έχουμε αυτοαπασχολούμενους. Χορτολιβαδικά είναι περίπου το 90% και το υπόλοιπο είναι καλλιέργειες. Αυτό εξηγεί πολλά πράγματα όσον αφορά τους κινδύνους του επαγγέλματος στην Ιρλανδία. Οι γεωργοί εργάζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ σκληρά και πολλές φορές δεν ανταμείβονται σωστά. Επίσης ε, εργάζονται στα αγροκτήματα ή τουλάχιστον επαροντες και μέλη της οικογένειας των γεωργών, όπως για παράδειγμα ηλικιωμένοι παιδιά. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι 400.000 άτομα είναι εκτεθειμένα σε διάφορες δύσκολες συνθήκες στα αγροκτήματα στις ουρικές εκμεταλλεύσεις Ιρλανδίας. Βλέπετε εδώ πέρα δύο γραφικές παραστάσεις, οι οποίες δείχνουν κάποιες μονάδες γαλακτοκομικών προϊόντων. Αριστερά έχετε τα εργατικά ατυχήματα, θανατηφόρα ατυχήματα και από την άλλη βλέπετε την ένταση των ατυχημάτων αυτών. Ουσιαστικά πάρα πολύ συχνά βλέπετε ότι όσο πιο εντατικό είναι το ατύχημα, όσο πιο σημαντικό είναι, τόσο πιο συχνά τελικά καταλήγει να είναι θανατηφόρο. εξετάζω το ζήτημα της ασφάλειας της γεωργίας σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούμε να πούμε ότι τα ποσοστά είναι πάνω κάτω τα ίδια. Αν κάνουμε μία γραφική παράσταση, ουσιαστικά θα δείχνει ίδια αποτελέσματα. Και ουσιαστικά, αν δούμε το ίδιο γράφημα για την Ιρλανδία, βλέπουμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια οι τάσει είναι ίδιε. Έχουμε δηλαδή μια επανάληψη των ίδιων ατυχημάτων. Ατυχήματα τα οποία βλέπουμε και στι άλλε χώρε. Στην Ιρλανδία εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι το ίμιση, το ίμιση των ατυχημάτων πλήττει άτομα που είναι άνω των 65 ετών. Και βλέπετε από τη γραφική παράσταση εδώ πέρα ότι ένα 70% θανατηφόρων ατυχημάτων συμβαίνουν σε άτομα άνω των 65 ετών. Άρα υπάρχει και ένα ηλικιακό παράγοντα πολύ σημαντικό. Τα θανατηφόρα αυτά ατυχήματα όμω είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου. Αν πάρουμε την περίπτωση των σοβαρών τραυματισμών, έχουμε ανθρώπου οι οποίοι τραυματίζονται πάρα πολύ σοβαρά, άνθρωποι που μένουν ανάπηροι και υπάρχουν ε, χιλιάδες γεωργοί οι οποίοι καταλήγουν σε αναπηρικά καρότσια κάθε χρόνο. Έχουμε μια εταιρική σχέση για την ασφάλεια στον τομέα της γεωργίας στην Ιρλανδία, ουσιαστικά ένας κοινωνικός διάλογος στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Έχουμε μάλιστα και ένα σχέδιο δράσης με 7 ομάδες εργασίας από 7 επαγγελματικούς τομείς που καλύπτει την περίοδο 2009 έως 2012. Έχουμε ένα σχέδιο προστασίας ε, της ε, ζωής, ε, της εργασίας μάλλον στη Γεωργία και έχουμε επίσης και έναν οδηγό ο οποίος περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία και υπάρχει ακόμα και ένα DVD με κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Επίσης στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δείτε κάποια άλλα εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς χρησιμοποιώντα απλώ το email του το password και να έχει μια καλύτερη καθοδήγηση όσον αφορά μια ασφαλή εξάσκηση του επαγγέλματο του Γεωργού. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε όλα αυτά τα DVD τα οποία καλύπτουν διάφορου τομεί. Το ζωικό κεφάλαιο, την γεωργική εκμετάλλευση, τα παιδιά στην γεωργική εκμετάλλευση και το Βέβαια τα προβλήματα εξακολουθούν και παραμένουν. Ακόμα και με όλου αυτούς τους οδηγούς και με όλα αυτά τα εργαλεία τελικά έχουμε ένα άτομο το οποίο χάνει κάθε δύο εβδομάδες τη ζωή του από κάποιο ατύχημα στη γεωργική εκμετάλλευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αλλάξουμε την οτροπία μας. Κάναμε μια πολύ σημαντική εκστρατεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου ε, λέγαμε στους ανθρώπους ότι δεν θα πρέπει να διακινδυνεύουν, πήγαμε σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια, δείξαμε την περίπτωση ενός ε, γεωργού ο οποίος χρησιμοποιώντας κάποιο γεωργικό μηχάνημα έχασε το χέρι του και ουσιαστικά θέλοντας να καταδείξουμε τα παραδείγματα αυτά θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Έγινε μάλιστα και μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο η οποία είναι αν θέλετε πάρα πολύ εντυπωσιακή, ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ακούγεται εκείνη τη στιγμή να υποφέρει κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, χρησιμοποιώντας μια μηχανή. Χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα μέσα, είναι διαθέσιμο όπως σας είπα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο, αλλά εξακολουθούμε και έχουμε πολλά προβλήματα ακόμα. Μολονότι οι γεωργοί στην Ιρλανδία προσπαθούν να εργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ουσιαστικά καταβάλουν πάρα πολλέ προσπάθειε προκειμένου να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο το ζήτημα τη ασφάλεια. Βλέπετε εδώ πέρα μία φωτογραφία ενός τρακτέρ το οποίο δεν περιέχει τις απαραίτητες, τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό που θα έπρεπε να έχει. Βλέπετε στη φωτογραφία αυτή ότι σε ένα σημείο χρησιμοποιείται απλώς ένα κομμάτι ξύλο αντί της βαλβίδας που θα έπρεπε να υπάρχει στο τρακτέρ αυτό και βλέπετε ότι τα μηχανήματα αυτά μπορούν να αποβούν πάρα πολύ επικίνδυνα. Για παράδειγμα βλέπετε εδώ πέρα μία οροφή, μία στέγη από την οποία έπεσε ένας γεωργός ηλικίας 70 ετών. Και βλέπετε εδώ πέρα κάποιον άλλον ο οποίος τραυματίστηκε πέφτοντας μέσα σε μία ανοιχτή δεξαμενή. Και βλέπετε εδώ πέρα στη φωτογραφία αυτή μία μάσκα οξυγόνου που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή ένα γεωργό προκειμένου να παραμείνει στην, στη ζωή μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Εδώ πέρα βλέπετε μία φωτογραφία ενό γεωργού ο οποίο οδήγησε με το τρακτέρ του πάνω στο παιδί του δύο ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα θνατηφόρων ατυχημάτων. Υπάρχουν περίοδοι οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από τόσο έντονο ποσοστό ατυχημάτων, αλλά επιστρέφουμε πάλι σε περιόδους με θανατηφόρα ατυχήματα. Προσπαθούμε να αναλύσουμε όλα αυτά τα δεδομένα στην Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία εργάζομαι και προσπαθούμε να δούμε σε πενταετή βάση ακριβώς τι γίνεται. Προσπαθούμε να αποκλείσουμε τον παράγοντα τύχη. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι μολονότι έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την κατάσταση τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, μολονότι έχουμε χρησιμοποιήσει όλο αυτό το διαφημιστικό υλικό, συνεχίζουν και αυξάνονται τα θανατηφόρα ατυχήματα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι απλώς πρόβλημα της Ιρλανδίας, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Θανατηφόρα ατυχήματα συμβαίνουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 574 είναι οι θάνατοι ετησίως κατά μέσο όρο και έχω μόνο δεδομένα από 12 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα μόνο για το 2007. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες, δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα επικαιροποιημένα, προκειμένου να καταφέρουμε να δούμε πώ έχει το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η Ιρλανδία έχει 15 θανάτους ανά 100.000, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχουν 9 εκατομμύρια, 9 θανάτους 100.000, στο Ηνωμένο, ε, μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 30. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια απόκληση στα δεδομένα αυτά. Πρέπει να ανταποκριθούμε στη Γεωργία σε όλες τις διαφορετικές πτυχές της, είτε είναι οικονομική αυτή, είτε είναι εμπορική, είτε είναι κοινωνική πτυχή. Υπάρχουν πολλά εκατομμύρια πολιτών που απασχολούνται στον τομέα της Γεωργίας και τη δασοκομεία επίσης. Όλοι γνωρίζουμε τα σημαντικά αυτά δεδομένα, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι τα άλλα δεδομένα. Το ότι έχουμε δηλαδή 600 θανάτους στον τομέα της γεωργίας σε αιτήσια βάση. Και ενδεχομένως τα πραγματικά δεδομένα να ανταποκρίνονται περισσότερο σε χίλια άτομα ετησίως. Όπω σα είπα, είχαμε δεδομένα από ορισμένα κράτη-μέλη μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο σίγουρο είναι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και επομένω χρειαζόμαστε μια πανευρωπαϊκή λύση. Θα πρέπει να έχουμε στρατηγικές για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, οι οποίες να λειτουργούν επί τόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η γεωργία να καλύπτεται από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να ισχύουν για άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Η στρατηγική ασφάλειας και υγείας συνεργασία, η κοινοτική και όλες οι σχετικές οδηγίες δεν εφαρμόζονται άμεσα σε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες όπως είναι για παράδειγμα οι η αλής, η η οι κτηνοτρόφοι. Θα δούμε τώρα την κοινή γεωργική πολιτική και τι διαπραγματεύσει που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Πραγματικά σκέφτομαι ότι ενδεχομένω να μπορέσουμε να βρούμε και κάποιε λύσει. Ενδεχομένω οι άμεσε ενισχύσει προ τα αγροκτήματα να μπορούν να συνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Δεν λέω ότι η απάντηση θα δοθεί μέσω των ενισχύσεων αυτών. Ενδεχομένω αν υπήρχαν άλλα προγράμματα, αν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα κατάρτισης, καλύτερης χρήσης των μηχανημάτων, αν υπήρχαν ε, οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας σε επίπεδο γεωρικής εκμετάλλευσης, ενδεχομένως τα πράγματα ήταν εντελώ διαφορετικά. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι εξίσου σημαντική με την καλή διαβίωση των ζώων, την βιοπικιλότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος. Κάνω λοιπόν μια, μια έκκληση προς εσάς σήμερα, προκειμένου η πολιτική υφιστάμενη να τροποποιηθεί. Οι υφιστάμενες στρατηγικές δεν αποδίδουν αποτελέσματα, δεν μπορώ να δώσω εγώ μια απάντηση, αλλά πρέπει μαζί να ψάξουμε για την καλύτερη λύση. Και δεχομένω να σφανεί λίγο περίεργο, αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να τρέφουμε την Ευρώπη μέσω της γεωργικής παραγωγής με ένα τίμημα σε πάρα πολλές ζωές Ευρωπαίων γεωργών που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Πέδρο Δελγάτο Κόμπος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή τη δημόσια ακρόαση εκ μέρους της Ένωσης Μικροκαλλιεργητών, Μικρογεωργών και Κτηνοτρόφων. Θα σας παρουσιάσω τις δραστηριότητες που πραγματοποιούμε στην Ισπανία υπέρ της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων και θα υποβάλω και κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, προτάσεις που επεξεργάστηκε η αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται. Θα ήθελα να σα πω ότι στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουμε στήσει μια Εθνική Επιτροπή Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με μια ομάδα εργασία που επικεντρώνεται στα προβλήματα του γεωργικού κλάδου. Επίσης, το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία, το οποίο ανήκω, ασχολείται ιδιαίτερα με τις εργασιακές συνθήκες στη Γεωργία. Έχουμε μάλιστα και μια δικτυακή πύλη για, το, για τη Γεωργία στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε και ένα εθνικό παρατηρητήριο για τις εργασιακές συνθήκες και εκεί έχουμε τα πορίσματα όλων των εθνικών ερευνών για τις εργασιακές συνθήκες. Εκεί συγκρίνουμε τα εργασιακά ατυχήματα στους διάφορους τομείς και ταυτόχρονα έχουμε και τα αποτελέσματα μιας εθνικής έρευνας που έχει γίνει ειδικά για τη γεωργία. Στις, μάλιστα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας και όλες τις μελέτες και τις έρευνες ε, σχετικά με το θέμα αυτό. Και θα σας αναφέρω τις προτάσεις της Εθνικής Αυτής Επιτροπής ε, για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η υγεία στη Γεωργία. Αυτή η Εθνική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι ένα συλλογικό όργανο που παρέχει συμβουλέ στι εθνικέ αρχέ για την διαμόρφωση πολιτικών, την πρόληψη και αποτελεί το θεσμικό όργανο συμμετοχή σε θέματα επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου μα ε, βλέπετε ποιο είναι το έργο αυτής της ομάδας για τη Γεωργία ειδικά και εκεί μπορείτε να ε, συμβουλευτείτε όλα τα έγγραφα εργασίας μας. Η Εθνική αυτή Επιτροπή απαρτίζεται από τέσσερις φορείς, από εκπροσώπους της ε, κεντρικής διοίκησης, από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους των εργοδοτών, των ε, επιχειρηματιών και εκπροσώπους των εργαζομένων. Και μάλιστα συντονιστικό όργανο είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας ε, στην Εργασία. Εκτός από την ομάδα εργασίας έχουμε και διάφορες υποομάδες, για παράδειγμα εποπτεία σε θέματα υγείας, ε, γεωργικά μηχανήματα, έχουμε υποομάδα για τα φυτογεωνομικά προϊόντα, για τα ζανιοκτώνα, ε, για, το, για τις εργασίες σε θερμοκήπια, γιατί στην Αλμερία, για παράδειγμα, έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και πυκνότητα ε, θερμοκηπίων. Έχουμε άλλη υπομάδα για την κτηνοτροφία, ε, μια υπομάδα για την ε, δασοκομεία, για την κατάρτιση και την ε, ενημέρωση, για το, το βαθμό των ατυχημάτων, τη εφαρμογή του νόμου σε ό,τι αφορά την αποτροπή των εργασιακών κινδύνων, για τις πυρκαγιές στα δάση και για τη διάσταση του φύλου έχουμε όλες αυτές τις υπομάδες που ανάλογα με τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις ανάγκες ε, ενεργοποιούνται και ε, αναλύουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης έχουμε μία ανάλυση των κινδύνων για κάθε θέμα. Εξετάζουμε τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν και εντοπίζουμε τις αδυναμίες, τα κενά των νομοθετικών διατάξεων, προτείνοντας κάποιες λύσεις. Στη συνέχεια έχουμε και πιο συγκεκριμένες προτάσεις για επιμέρους προβλήματα. Μάλιστα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου μας μπορείτε να εξετάσετε όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένα link με το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Εργασιακές Ηθίκες, με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας και επίσης ένα σύνδεσμο για, με τις θεματικές δικτυακές πύλες. Μια δικτυακή πύλη ε, ειδική για τη γεωργία. Εδώ είναι η ιστοσελίδα μα για τη γεωργία με διάφορε υποκατηγορίε για τα γεωργικά μηχανήματα, για τα φυτογειονομικά προϊόντα, για τι δασοκομικέ δραστηριότητε, ε, κτηνοτροφία και ούτω καθεξής. Επίσης, σε αυτή την ιστοσελίδα έχετε πρόσβαση και στο Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Εργασιακές Συνθήκες. Εκεί περιλαμβάνουμε τα απορίσματα όλων των εθνικών μελετών και ερευνών που αφορούν τις εργασιακέ συνθήκες. Στην τελευταία εθνική απογραφή και έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες το 2012 θα ήθελα να σας αναφέρω τη σύγκριση που γίνεται μεταξύ των διαφόρων τομέων της γεωργίας, της βιομηχανίας, του κατασκευαστικού κλάδου και των υπηρεσιών. Και βλέπουμε τη την σημασία που έχουν κάποιες ε, μυοσκελετικές ε, διαταραχές ή προβλήματα ανάλογα με το που απασχολείται ο καθένας. Και εδώ έχουμε την σελίδα από μια εθνική έκθεση σε ό,τι αφορά την αγροπιστιστικό κλάδο. Ε, ταυτόχρονα γίνονται διάφορες έρευνες για τις εργασίες, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις δονήσεις στη γεωργία. Είναι ένα από τα προβλήματα που τελευταία ανέκυψαν και αφορούν πάλι κάποια μειοσκελετικά προβλήματα εξαιτία των δονήσεων. Δεν θα επεκταθώ. Θα ήθελα να περάσω στις τελευταίες μου διαφάνειες. Από τις διάφορες υπομάδες που σας παρουσίασα, συγκεντρώσαμε προτάσεις που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητες ε, όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλες χώρες. Η πρώτη πρόταση αφορά την προώθηση της ε, εκπόνησης ειδική ε, νομοθεσίας για την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων στη Γεωργία. Γνωρίζουμε ότι έγινε μια απόπειρα δημοσίευσης ή εκπόνησης μιας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη Γεωργία, αλλά δυστυχώς δεν ευωδόθηκαν αυτές οι προσπάθειες. Πρόσφατα όμως είχαμε τον Ευρωπαϊκό Οδηγό, το Ευρωπαϊκό Χειρίδιο για την Γεωργία, αλλά δυστυχώς για μας στην Ισπανία ε, δεν υπάρχει ο οδηγός αυτός μεταφρασμένος στα ισπανικά. Αρχικά είχε προβλεφθεί η μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς πρόσφατα έμαθα ότι μόνο σε μια γλώσσα, μόνο σε λίγες γλώσσες κυκλοφορεί αυτός ο οδηγός, μόνο στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση να προσπαθήσετε, αν γίνεται, να μεταφράσετε και στα Ισπανικά αυτόν τον οδηγό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μα. Δεύτερη πρόταση που προέκυψε από αυτέ τι υποομάδε. Η ενίσχυση και προώθηση ε, των, ε, της πρόληψης, ιδιαίτερα στη Γεωργία. Η πρόληψη των κινδύνων στις επιχειρήσεις ε, στην Ισπανία γίνεται κυρίως μέσω κάποιων υπηρεσιών πρόληψης αλλά που όμως είναι πολύ ασήμαντες, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα της πρόληψης. Δεν έχουμε. Συνήθως είναι ξένες, είναι εξωτερικές της γεωργίας αυτές οι υπηρεσίες πρόληψης. Θα πρέπει ο ίδιος ο γεωργός να προσλάβει κάποιον που να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Θέλουμε όμως ένα κοινό φορέα που να ασχολείται με την πρόληψη κινδύνου στη γεωργία και να μπορούν σε αυτό να έχουν πρόσβαση πολύ περισσότεροι γεωργοί. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος αυτών των υπηρεσιών πρόληψης. Μία άλλη πρόταση αφορά την διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατιών για την ενημέρωση, κατάρτιση και συνειδητοποίηση των κινδύνων της γεωργίας με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, στους αυτοπασχολούμενους και τους αυτόνομους εργαζόμενους. Θέλουμε διεξαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων των γεωργικών ε, μηχανημάτων και σε ό,τι αφορά τη θέση του σε εμπορία και τη χρήση, άσχετα με το είδος του χρήστη. Συνήθως οι προδιαγραφές αυτών των γεωργικών μηχανημάτων είναι διαφορετικές ε, ανάλογα με το αν ο εργαζόμενος είναι αυτόνομος ή εργαζόμενος, μισθωτός για τον αυτόνομο απαιτείται περισσότερη ασφάλεια. Θεωρούμε ότι οι ψηλέ προδιαγραφέ ασφάλεια θα πρέπει να ισχύουν για όλου, άσχετα με το είδο τη εργασιακή σχέση. Άλλη πρόταση αφορά την πρόθεση ε, κάποιων, ε, απαραίτ, κάποιων ε, απαραίτητων προδιαγραφών κατάρτισης για όσους χειρίζονται συγκεκριμένα μηχανήματα όπως είναι ε, μετατοπιστές, αλυσοπρίωνα, μεταποιητές και ούτω καθεξής καθώς και μια ομοιογενοποίηση της κατάρτισης σε, σε τέτοια θέματα και θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ώστε να υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης στις διάφορες περιοχές. Άλλη πρότασή μας αφορά την ανάπτυξη και ε, μάλλον την εκπόνηση και ε, διάδοση χειριδίων βέλτιστων πρακτικών για την ασφαλή ε, χρήση των γεωργικών μηχανημάτων που περιλαμβάνει τους απαραίτητους ελέγχους, τεχνικούς ελέγχους και τον τρόπο συντήρησης αυτών των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και τον οδηγό με, με, καθώς και τις οδηγίες χρήσης και φυσικά πρόθεση των μελετών, προσαρμογή και βελτίωση των εξοπλισμών και των τεχνικών εφαρμογής, προς, προώθηση της ε, προσαρμογής και βελτίωσης της, ε, των προσωπικού, μηχανισμού προστασίας και φυσικά ε, να γενικεύσουμε την, την πρόληψη στη γεωργία και την να επαγρυπνούμε για την εξασφάλιση της υγείας και της προστασίας. Εδώ έχουμε ένα καροτσάκι για το ψεκασμό σε, θερμοκήπια. Και εδώ έχουμε ένα, ε, μια, ε, ε, ένα τόξο ασφάλειας που αυτόματα ενεργοποιείται σε περίπτωση που το όχημα, ελκυστήρας, αποκτήσει μια συγκεκριμένη κλίση. Πάνω από την κλίση αυτή ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός προστασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές και τώρα καλώ τον πρόεδρο κύριο Μάνα να κάνει την παρουσίαση των άλλων ομιλητών. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι. Μπορώ να σας παρουσιάσω το προσεχή ομιλητή, τον Πολ Γάλλο. Έχει ετοιμάσει ένα σημείωμα. Σας το διαβάζω στο αγγλικά. Είναι γεωργός από την Νότια Γαλλία. Έχει ιδρύσει ένα κίνημα μεταξύ των γεωργών βιομηχανικού της έκτασης και ιατρών στην περιοχή του και αυτό ύστερα από έκθεση και συνέπειες στην υγεία του ε, κατά τη διάρκεια της εργασίας του για να αγωνίστηκε για να αναγνωριστεί ως επαγγελματική ασθένεια. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος της πράξης και περιμένουμε να τον ακούσουμε για να ε, μας περιγράψει την εμπειρία του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, ε, μιλάω μόνο γαλλικά. Είμαι γεωργός και πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι δέος που βρίσκομαι σε τέτοιο ακροατήριο. Θα σας ε, παρουσιάσω την ε, γεωργία μας, την οργάνωσή μας και τις εμπειρίες μας. Πρόκειται για μια οργάνωση την οποία ιδρύσαμε ε, όταν διαπιστώσαμε πριν από δύο χρόνια Ε, διότι με το σχέδιο που ξεκίνησα διαπίστωσα ότι υπήρχαν και άλλοι ε, γεωργοί που είχαν υποστεί δηλητηρίαση από τα γεωργικά προϊόντα και έτσι διαπιστώσαμε ότι ήταν αναγκαίο να συνεργαστούμε ώστε καταρχάς να πάψει η σιωπή των γεωργών γιατί είναι δύσκολο να, γνωριστεί, ε, να αναγνωρίσει κάποιος ότι μπορεί να εάν αρρώσει γι' αυτό να είναι υπέτειο στο τρόπο του, το επάγγελμά του. Φτιάξαμε λοιπόν αυτήν την οργάνωση και χάρη σε αυτήν ε, και είπαμε ότι χρειάζεται να βελτιωθεί η αναγνώριση των ε, φυτογειονομικών προϊόντων και γιατί να θα αναφερθώ στα αυτά που είδαμε νωρίτερα για τα ατυχήματα στην Ιρλανδία. Πολύ λίγοι αναφορά γίνεται ε, στα προβλήματα υγείας που εμφανίζονται από τη χρήση χημικών ουσιών στη γεωργία και όμως όλο και πιο πολύ αναγνωρίζεται ότι οι καρκίνοι οφείλονται σε εξωτερική ρήπανση. Η Γαλλία που καταναλώνει και πολλά γεωργικά προϊόντα, με συγχωρείτε με κάπως ταραγμένος, ε, Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την αναγνώριση της επαγγελματικής ασθένειας καταρχάς, γιατί αυτό επιτρέπει καταρχάς την κάλυψη από τις κοινωνικές υπηρεσίες του ασθενούς. Αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στη Γαλλία, δεν αναγνωρίζεται η ειδική γεωργική ε, από την ειδική γεωργική εταιρεία ασφάλισης ε, η επαγγελματική νόσος πλην της Πάρκινσον ως ε, νόσου που προξενούν τα ε, φυτοφάρμακα και μόνο ε, το φυτοφάρμακο που αποτελεί ένωση του αρσενικού αναγνωρίζεται ως επικίνδυνο από την εν λόγω αλληλεσφαριστική εταιρεία. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος δεν γνωρίζει πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το προϊόν του. Επίσης, δε, ε, θεωρούν πολλοί γεωργοί ότι δεν έχουν συνέπειε στην ε, υγεία τους οι ε, ουσίες που χρησιμοποιούν. Γιατί εγώ μπορεί να πέσω θύμα μιας οξίας δηλητηρίασης, αλλά οι περισσότεροι πάσχουν από χρόνια δηλητηρίαση. Μέσα σε 30 χρόνια περίπου μπορεί να εμφανιστεί η παθολογία την οποία έχουν προξενήσει οι ουσίες που χρησιμοποιούν στην γεωργία. Και γιατί ζητούμε να βελτιωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η παρακολούθηση και η χνηλασιμότητα των προϊόντων. Στη Γαλλία έγινε μια ε, συνάντηση, ένα συνέδριο στην Νότια της Γαλλίας όπου ε, προβλήθηκε και τις δημόσιες υπηρεσίες ότι υποτιμάται η σημασία και η βαρύτητα των ε, χημικών ουσιών χρησιμοποιούνται στη Γεωργία. Επίσης από την Γερουσία της Γαλλίας ε, εκδόθηκε μια έκθεση που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2012 ε, με υπογραφές από όλους τους βουλευτές, όλο, από τους βουλευτές όλων των κομμάτων που καταδεικνύει ακριβώς τους κινδύνους και για τους περίγους και για τους γεωργούς αλλά και για τους καταναλωτές των γεωργικών προϊόντων. Υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν ε, χρηματοδοτήσει μελέτες, όχι ακριβώς μελέτες, μάλιστα μια έρευνα είναι μόνο, που καταγράφει τις συνέπειες ως προς τον γεωργό, την υγεία του, τον Την υγεία του περίοικου. Και είναι κρίμα το ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι αυτέ που αναλαμβάνουν τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Εμεί, η Ένωσή μα δηλαδή, αγωνιζόμαστε ώστε οι κρατικέ υπηρεσίε να αναλάβουν τις ευθύνε τους, γιατί ορισμένοι μας κατηγορούν ε, για η δραματοποίηση της κατάστασης, για παρουσίαση της κατάστασης τραγικής, αλλά εμεί αυτό που ζητούμε είναι να διατεθούν περισσότερα κονδύλια, γιατί χρήματα πάντα χρειάζονται, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο περιθώριο για αβεβαιότητα. Η εναρμόνιση επίση έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Ε, δίπλα μου κάθε ένας Ισπανός. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προϊόντα απαγορευμένα στη Γαλλία, που κυκλοφορούν ελεύθερα στη Γαλλία. Ή το αντίστροφο. Και Ζητώ συγγνώμη αν μιλάω κάπως ομά. Υπάρχει περίπτωση, ή πάντως μας, ε, μας απασχολεί το εάν υπάρχουν ε, μεγάλες εταιρείες οι οποίες ε, αποδέχονται την απαγόρευση ενό προϊόντος σε μία χώρα, προκειμένου να μπορούν να το παραγάγουν και να του επιτρέψουν κυκλοφορία, να το διαθέσουν αγορά ελεύθερα σε μία άλλη και να λειτουργήσουν με βάση τι παράλληλε ε, εξαγωγέ. Δηλαδή από την Ισπανία ένα προϊόν που είναι απαγορευμένο στη Γαλλία να έρχεται στην επικράτειά μα ε, χωρί έλεγχο. Επίση πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλοί γεωργοί που εργάζονται χωρί καμία προληπτική δράση. Το είδαμε και από τις παρουσιάσεις. Βεβαίως το μηχανολογικό σκέλος είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά από την άλλη με ε, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά σε όλους αυτούς τους γεωργούς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες αυτή τη στιγμή και δεν καταγράφονται στατιστικές. Εμείς βλέπουμε ότι είναι πολλοί οι γεωργοί μεταξύ 40 και 45 και ιδιαίτερα στο ναμπελοϊνικό τομέα που έχουν ε, παρουσιάσει καρκίνου της ηροδόχου κίστης, των όρχεων, του προστάτη και αντίστοιχες ε, παθήσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία εμείς από κοντά να το εξετάσουμε και για τις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης. Ε, στη, στη Ρουμανία, την οποία επισκέφθηκα μόλις αυτό το Σαββατοκυριακό και δεν σας μιλάω για τον τρόπο που εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν μιλάμε ούτε για ε, συνέπειες στην υγεία τους, προϊόντων που χειρίζονται με γυμνά χέρια γιατί κανείς δεν τους έχει μιλήσει για προστασία ε, και προστατευτικό εξοπλισμό. Θα δούμε σε μερικά χρόνια ποια θα είναι η κατάσταση τη του. Τώρα, ό,τι και να μα πούν οι Γάλλοι πολιτικοί, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν ήταν ενήμεροι. Η κατάσταση είναι τραγική. Οι γεωργοί ε, λένε «Αχ, έχω 400 εκτάρια, είναι αρκετά μεγάλη εκμεταλλευσή μου, δεν θεωρούμε βιολογικός γεωργός, χρησιμοποιώ τα χημικά ε, προϊόντα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο πριν, αλλά, αλλά τα γεωργικά προϊόντα πλέον δεν είναι απαραίτητα στη γεωργία και αν, μπορεί κανείς να αν ε, θέλει κανείς να ισχυριστεί ότι μπορεί η γεωργία να κινδυνεύσει στην Ευρώπη με τον περιορισμό της χρήσης των χημικών ουσιών, είναι ψέμα, είναι σφάλμα, σας διαβεβαιώνω ότι γίνεται να ζήσει κανεί και φαντάζομαι ότι θα καταλάβετε τον τρόπο που εκφράζομαι ότι δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ένα απλό γεωργό. Γίνεται να επιβιώσει κανεί μόνο με τη γεωργική δραστηριότητα χωρί αυτά τα προϊόντα. Και ήθελα στην κατάληξή μου να πω ότι χρειάζεται να έχουμε μια παραγωγή καθαρή που να σέβεται το περιβάλλον, που να προάγει ε, τι αγρονομικέ ε, αρχέ και το σεβασμό του περιβάλλοντο, ανάλογα με τι συνθήκε που επικρατούν στην κάθε περιοχή, γιατί οτιδήποτε μπορεί να πω ότι ισχύει για τη δική μου την περιοχή δεν ισχύει απαραίτητα και στη Γερμανία ή στην Ισπανία ή σε κάποια γειτονιά, σε κάποια περιοχή της Ιταλίας. Αλλά οτιδήποτε γίνει, οτιδήποτε κακό και λάθος γίνει στην ε, ύπεθρό μας, στα, ε, στα χωράφια μας, θα έχει συνέπειες για ολόκληρη την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. Και ευχαριστώντας σας, θα ήθελα να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη για τα πολλά λάθη στην γλώσσα που έκανα. Monsieur also ich habe kein... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λεφόνσο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ελπίζω ότι αισθάνεστε κι εσείς άνετα σε αυτό το αμφί, όπως το λέτε, τόσο ωραία το αμφιθέατρο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν κοιτάμε κανένα αμφιψηλού, ότι σεβόμαστε κάθε παρουσία εδώ και ότι θέλουμε να δούμε όλα τα προβλήματα σε κάθε σημείο και θέλουμε πάνω απ' όλα κάθε γεωργός να γνωρίζει όταν χειρίζεται μια ουσία τι είδους συνέπειες μπορεί αυτή να έχει. Και θέλουμε ε, και οι υπηρεσίες να δείξουν ε, την αναλυτική πλευρά της δουλειάς τους. Η κυρία Πλόνιτσε που είναι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Υγεία και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Την περιμένουμε με αδημονία για να ακούσουμε την ανάλυση της με τις βασικές ιδέες και με πρακτικά παραδείγματα. Έχετε το λόγο. Uh, thank Ευχαριστώ. Θα σας κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή των χαρακτηριστικών του κλάδου και θα σας παρουσιάσω τις προσπάθειες της, του δικού μου οργανισμού για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της γεωργίας και θα αναφέρω για κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Ο γεωργικός κλάδος είναι μικρός αλλά σημαντικός. Το 5% ε, απασχολείται στην Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριαρχείται από άνδρες, το 65%. Ε, είναι χαμηλά σχετικά τα μορφωτικά επίπεδα, ε, η ανειδίκευτη επίση εργασία είναι υψηλή και το εισόδημα των γεωργών δυστυχώς χαμηλό. Οι περισσότεροι γεωργοί είναι αυτοαπασχολούμενοι. Το 78% μόνο, απασχολείται μόνο του και είναι μεγάλο, το από μάλλον απασχολείται το 78% εργάζονται μόνοι τους ή με τη βοήθεια των μελών της οικογένειάς τους και οι περισσότεροι είναι εποχικοί εργαζόμενοι. Τα, οι προσωρινές συμβάσεις φτάνουν στο 43,9%, 24% δεν έχουν καν κάποιο συμβόλαιο και οι περισσότεροι είναι μετανάστες. Σας τα αναφέρω όλα αυτά γιατί τα χαρακτηριστικά της γεωργίας έχουν ε, επίπτωση στην ε, ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την, το σχεδιασμό προτάσεων και την ανάληψη νέων πρωτοβουλειών για την διόρθωση των προβλημάτων. Πολλές είναι οι δραστηριότητες στο γεωργικό κλάδο και διαφορετική είναι και η κίνδυνη για την υγεία. Θα αναφερθώ σε ορισμένα μόνο παραδείγματα. ακούσαμε κάποια εργασιακά ατυχήματα, αλλά για τους νέους εργαζόμενους το μεγαλύτερο η μεγαλύτερη το μεγαλύτερο ποσοστό ε, θανατηφόρων εργασιακών ατυχημάτων εντοπίζεται στη Γεωργία. Σε ό,τι αφορά τους ε, κινδύνους για, τη, την υγεία, είναι εργονομική, ε, θέματα χορύπανσης, δόνησης, η εργασία σε ψυχρό ή υπερβολικά θερμοπεριβάλλον, η χρήση των φυτοφαρμάκων και παρασιτοκτόνων. Επίσης μπορεί να έχουμε οξύς, δηλητηριάση εξαιτία των φυτοφαρμάκων, αλλά έχουμε και χρόνια μακροπρόθεσμα προβλήματα στην υγεία που δεν αναγνωρίζονται δυστυχώ ε, ε, ως, εργασιακή κίνδυνη. Για παράδειγμα, εξαιτία της χρήσης φυτοφαρμάκων μπορούν να αναπτυχθούν ε, καρκίνοι, πάρκινσον, προβλήματα στη γονιμότητα, προβλήματα στην αναπαραγωγική υγεία, ακόμη και κατάθλιψη και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη τα ατυχήματα και τους κινδύνους, ε, πολλές φορές ε, δεν λαμβάνουμε υπόψη τους ε, ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τους κινδύνους για την πνευματική υγεία, την ψυχική υγεία. Με βάση έρευνες διαπιστώνουμε υψηλά επίπεδα τέτοιου είδους κινδύνων, για παράδειγμα μεγάλες παρατεταμένα ωραία εργασίας, δυστυχώς μη ισορροπημένη ε, ζωή, ε, λίγες κοινωνικές επαφές, ε, ελάχιστες προοπτικές σταδιοδρομίας και σε με την υγεία προβλήματα, άγχος, στρες, διαταραχές του ύπνου, μεγάλη κόπωση και μεγάλο ποσοστό εργαζομένων παραπονούνται για κακή ψυχική υγεία και μάλιστα 40% των γυναικών και 22% των ανδρών που απασχολούνται στον κλάδο ε, εκφράζουν παράπονα για τέτοιου είδους προβλήματα. Πολλές είναι βέβαια και οι προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της ε, επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας ε, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτού του κλάδου. Πολλοί εργαζόμενοι δεν είναι καλά κατατοπισμένοι για τους κινδύνους ε, στην ασφάλεια και την υγεία. Μόνο το 20% των εργαζομένων ε, ε γνωρίζουν την ανάγκη κατάρτισης και επίσης υπάρχει χαμηλό επίπεδο εκπροσώπησης των εργαζομένων. Υπάρχουν και πολύ ισχυροί πολιτιστικοί και συμπεριφερολογικοί παράγοντες για παράδειγμα, πολλοί επικαλούνται την παράδοση. Έτσι έκανε ο παππούς μου, ο μπαμπάς μου και εγώ το ίδιο σε όλη μου τη ζωή. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να αλλάξω μια τέτοια συμπεριφορά. Δύσκολο είναι επίσης να ε, φτάσουμε σε όλους τους γεωργούς, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχουν πολύ μικρές καλλιέργειες και άλλη πλέον δηλαδή πρόκληση. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την υγεία και την προστασία, την ασφάλεια στη, Γεωργία. Καταρχήν θα πρέπει να αφυπνίσουμε τους ενδιαφερόμενους για τα προβλήματα και θα μπορούσαμε έτσι κυρίως να τους παρουσιάσουμε κάποια καθημερινά παραδείγματα. Πώς μπορούμε τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας να βελτιώσουν και την οικονομική διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης να τους ενημερώσουμε για παραδείγματα προς μίμηση αλλά και για παραδείγματα προς αποφυγή. Για το τι μπορεί να γίνει δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθήσει κανείς καλές πρακτικές υγείας και ασφάλειας. Επίσης θα μπορούμε να διαδίδουμε τις καλές πρακτικές και να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση γιατί Μπορεί ένα Γεωργό να μην ακούει τα κρατικά όργανα ή τι αρμόδιε αρχέ, αλλά πολύ εύκολα να ακούσει το γείτονα γεωργό. Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι γεωργοί υφίστανται πιέσει ε, και λόγω έλλειψη χρόνου και λόγω οικονομικών δυσχεριών. Γι' αυτό δεν έχουν το χρόνο να μεταβούν στην πρωτεύουσα σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο για να παρακολουθήσουν σεμινάριο. Οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε και με επιχειρήσεις που έχουν σχέση υπεργολαβίας με γεωργούς και να χρησιμοποιούμε φυσικά πρακτικούς ε, τρόπους αξιολόγηση του κινδύνου. Το σημαντικό όμω είναι να αλλάξει η νοοτροπία, να αλλάξει η συμπεριφορά των γεωργών και να αντιληφθεί ο γεωργός ότι η υγεία και η προστασία στην εργασία θα έχει θετικά αποτελέσματα και στην οικονομική διαχείριση και στην αποδοτικότητα της γεωργικής εκμετάλλευση. Ο οργανισμός μου έχει αναλάβει πολλές δραστηριότητες, κυρίως σε τρεις τομείς. Προσπαθούμε καταρχήν να αφυπνίσουμε τους ενδιαφερόμενους με αιτήσεις ενημερωτικές εκστρατείες, με διάφορα θέματα κάθε φορά. Είχαμε μια ενημερωτική εκστρατεία για τη γεωργία. Σε κάθε ενημερωτική εκστρατεία πάντως περιλαμβάνουμε και τη γεωργία ως κλάδο. Τώρα έχουμε την εκστρατεία συνεργασία για την πρόληψη του κινδύνου. Επίσης θέλουμε να διαδίδουμε τις καλές πρακτικές και έχουμε πολύ καλό παράδειγμα από την Ιρλανδία όπου 15 ε, ε, ε, συνεργάζονται και συνέρχονται κάθε μήνα προκειμένου να συζητούν τις διάφορες ε, βέλτιστες πρακτικές κτηνοτροφίας, αλλά ασχολούνται και με θέματα ασφάλειας και υγεία στην εργασία και μάλιστα χρησιμοποιούν και κάποια εργαλεία online για αξιολόγηση του κινδύνου και θεωρούν ότι τέτοια εργαλεία είναι πολύ χρήσιμα και πολύ προσετά. Επίσης εξετάζουν τους κινδύνου σε όλους τις εκμεταλλεύσεις και μας ε, δήλωσαν ότι θα ήταν χρήσιμο να ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο και άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και μάλιστα έτσι έχουν και ε, εξωτερικούς ε, παρατηρητές που είναι ε, πιο αμερόληπτοι και πιο ουδέτεροι. Γιατί όταν κανείς εργάζεται σε μια επιχείρηση, πολύ συχνά, επειδή ακριβώ το μάτι του κυκλώνα, δεν βλέπει τα προβλήματα. Ένας εξωτερικός παρατηρητής θα εντοπίζει καλύτερα. Επίσης, Έχουμε τη διάδοση των καλών πρακτικών με ε, συγκεκριμένη ανάλυση προβλημάτων, με χρήση των τεχνολογιών και του διαδικτύου, τις πιο συχνές ερωτήσεις, τη συλλογή των εργαλείων για εκτίμηση του κινδύνου και τη συντηρήση στη γεωργία με τον οδηγό μας. Επίσης, συλλογή δεδομένων έχουμε και την, ε, την, έκθεση, την ε, έρευνα που γίνεται στις επιχειρήσεις και στην τελευταία μας έρευνα περιέλαβαμε και τη γεωργία. Θα εξετάσουμε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από πέντε εργαζόμενους. Θα δούμε λοιπόν ε, ποιοι είναι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, οι εργασιακοί κίνδυνοι σε τέτοιου τους επιχειρήσεις και τώρα, με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την οργάνωση ημερίδων για την συνειδητοποίηση της υγείας και της προστασίας στην Γεωργία και εκεί έχουμε πρακτικά παραδείγματα και επιδείξεις σε ό,τι αφορά κινδύνους που κυρίως απειλούν τους εργαζόμενους στη Γεωργία ή τα μέλη των οικογενειών τους. Πάνω από 43.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, 140 τον αριθμό από, το, από τις ημερίδες αυτές για την ενημέρωση και ε, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι χάρη στι μερίδε αυτέ ε, κατάφεραν να ενσωματώσουν στη δική του γεωργική επιτάλευση τουλάχιστον ένα από του κανόνε για την ε, ασφάλεια και προστασία. Και μάλιστα όλοι όσοι συμμετείχαν και παρακολούθησαν αυτέ τι εκδηλώσει τι συστήνουν θερμά και στου υπόλοιπου γεωργού. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώ μπορούμε να φτάσουμε σε όλους τους γεωργούς. πληροφορίες, για περισσότερες πληροφορίες θα παραπέμπω στο, στην ιστοσελίδα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κύριος ε, ο κύριο Συμπρόεδρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές μας για όλες αυτέ τι παρουσιάσει. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Χέρπλεστον να μιλήσει εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να αναφερθώ σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον τομέα της γεωργίας. Μάθιου Χάλπιλτς ονομάζομαι, εργάζομαι για τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο, ιδίως για ζητήματα ασφάλειας και υγείας στον τομέα της εργασίας. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ευρωπαϊκές πολιτικές για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Επίσης, όπως είπαν και οι ομιλητές, βλέπουμε ότι το επίπεδο ασφάλειας και υγείας στη Γεωργία μας προκαλεί ανησυχίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τραυματίζονται, χάνουν τη ζωή τους με πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία. Βέβαια, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας, ωστόσο όμως υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Αν δούμε τώρα την κοινοτική στρατηγική από το 2007 μέχρι το 2012, προσπαθούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα εργατικά ατυχήματα καθώς επίσης και τις εργατικές ασθένειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα νομοθετήματα και πολιτικές που θα πρέπει να ενδυναμωθούν και θα πρέπει να επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίω σε κάποιους τομείς υψηλού κινδύνου όπως η γεωργία, η αλία, οι μεταφορές και ο κατασκευαστικό τομέα. Η στρατηγική επίση Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι κάποια παραδοσιακά μη δεσμευτικά μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να γίνουν κατανοητά από όλου, να συνειδητοποιήσουν όλοι ποιοι είναι οι υποχρεώσει του και θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέσα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται πολύ στενά με την Τριμερή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον χώρο της εργασίας και με όλου τους επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μη δεσμευτικός οδηγός. Ο οδηγό αυτό φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει όλου του εμπλεκόμενου στον τομέα τη γεωργία και τη αστυνομία, του ίδιου του γεωκτήμονε, του γεωργού, εργοδότες και εργαζόμενους, προκειμένου να καταφέρουμε να ελοποιήσουμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθηθούν κάποια θετικά παραδείγματα και κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εθνική νομοθεσία, γιατί ενδεχομένως σε εθνικό επίπεδο ορισμένα κράτη-μέλη να θέλουν να υιοθετήσουν πιο αυστηρά μέτρα από αυτά τα οποία προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία επιλέξαμε τελικά έναν μη δεσμευτικό οδηγό γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια κοινοτική οδηγία, νομοθεσία όσον αφορά τους εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας, κοινοτροφίας και της δασοκομείας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τομέων αυτών, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην Ήπεθρο με ζωικό κεφάλαιο χρησιμοποιώντας γεωργικά μηχανήματα πολλές φορές μόνοι τους απομονωμένοι με, χαμηλό επίπεδο, με χαμηλό χρησιμοποιώντας χημικά προϊόντα Όλοι αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν το προφίλ κινδύνου και οδηγούν σε περισσότερα ατυχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπώς αποφάσισε να εκπονήσει αυτό το μη δεσμευτικό οδηγό. Είναι ήδη διαθέσιμο σε 200 σελίδες και 21 κεφάλαια. Δίνει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και αναφέρεται επίσης και σε άλλα σημαντικά στοιχεία όπως κάποιες επεξηγήσεις για το πώς μπορεί να κάνει κανείς μια σωστή αξιολόγηση του κινδύνου κατά τη διάρκεια της γεωργικής δραστηριότητας. Ένα καινοτόμο στοιχείο το οποίο περιέχει ο οδηγό είναι το ότι χρησιμοποιείται ένα διαδραστικό μέσο αξιολόγηση του κινδύνου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο, μπορεί να εκ των προτέρων να κάνει ένα κατάλογο επικίνδυνων παραγόντων και να καταφέρει να συνειδητοποιήσει τελικά ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου το οποίο υφίσταται στη γεωργική του μονάδα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης κινδύνου που συνδέονται για παράδειγμα με το να μπορεί κανείς να επιλέξει τον επαγγελματικό του τομέα, γιατί βέβαια δεν έχουν όλοι οι τομείς τα ίδια χαρακτηριστικά, ή μπορεί κανείς να επιλέξει πιο συγκεκριμένα τη δραστηριότητα την οποία θέλει να αξιολογήσει και να κάνει έπειτα μια παραμετροποίηση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγελματικού κλάδου, τα οποία σας ανέφερα, και όπως σας είπα μπορεί κανείς ακόμα και σε επίπεδο γεωργική μονάδας να δημιουργήσει αν θέλετε λίγο το, το προφίλ επικινδυνότητας που μπορεί να έχει η γεωργική του εκμετάλλευση. Σε αυτόν τον τρόπο μπορεί κανεί να συνειδητοποιήσει ποια δράση πρέπει να λάβει και σε ποια χρονική στιγμή θα πρέπει να ληφθεί αυτή η δράση. Ωστόσο θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να είμαστε κάπω προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτού του οδηγού. Εφόσον κάθε χώρο εργασίας διαφέρει και κάθε επάγγελμα ουσιαστικά είναι διαφορετικό, οι συστάσει και οι προτάσει που γίνονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έναν απόλυτο κανόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογήσει πρώτα ο Γεωργό την υφιστάμενη κατάσταση στη γεωργική του μονάδα και να προσαρμόσει ουσιαστικά τον οδηγό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση ο Γεωργό να σέβεται και την εθνική νομοθεσία και τι εθνικέ προποθέσει που ισχύουν στο αγρόκτημά του με βάση τη χώρα στην οποία βρίσκεται. Εν κατακλείδη πρέπει να σας πω ότι ο οδηγός αυτός είναι διαθέσιμο σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Και ένα από τα ζητήματα που έχουμε εντοπίσει είναι να δούμε πώ θα καταφέρουμε τελικά να διανύμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οδηγό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι τελικοί αποδέκτε να καταφέρουν να λάβουν στα χέρια του τον οδηγό αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διανύμουμε τον οδηγό μέσω των εθνικών σημείων επαφή που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια αντίτυπα του οδηγού αυτού σήμερα στην αίθουσα αυτή. Εφόσον ενδιαφέρεστε, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Μπορεί να, μπορεί να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Οι ομιλητές έχουν δύο λεπτά στη διάθεσή τους και στη συνέχεια θα απαντήσουν οι πυρογνώμονες. Η κυρία Μογάν Σαχτιέ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας για τις πολύ κατατοπιστικές τους παρουσιάσεις και διαφωτιστικές εμπειρίες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Ό,τι μορφή γεωργίας και αν ασκούν. Α, βέβαια διαπιστώνουμε ότι σήμερα οι κίνδυνοι αυτοί εντείνονται γιατί πριν από 30 χρόνια για παράδειγμα οι γεωργοί μας ήταν αυτοί που είχαν το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Βλέπετε από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει σήμερα. Πού καταντήσαμε στην ουσία. Γιατί αν κάνουμε σύγκριση με το παρελθόν βλέπουμε ε, πόσο έχει υποβαθμιστεί η κατάσταση και τι επιτακτική ανάγκη υπάρχει για άμεση δράση. Πολύ καλή παρουσίαση ε, ενό τεράστιου φάσματο ε, κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Γεωργοί. Ο κύριο Φρανσουά ήταν ζωντανό παράδειγμα και υπάρχει μια κατηγορία κινδύνων που δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και μερικέ φορέ του παραμελούμε. Πολύ συχνά οι Γεωργοί βρίσκονται ε, σε κανονικούς δρόμους, κινούνται σε κανονικούς δρόμους ή αυτοκινητοδρόμους μαζί με οχήματα που έχουν διαφορετική ε, ταχύτητα και διαφορετικό είδος κίνησης. Αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο για τους γεωργούς. Δεν έχουν ε, δικούς τους περιφερειακούς επαρχιακούς δρόμους που μπορούν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά, αλλά χρειάζεται να κινούνται μέσω των εθνικών οδών μαζί με τα υπόλοιπα οχήματα ιδιωτικής ή άλλης χρήσης. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι διαπιστώνουμε την ανάγκη συνειδητοποίησης του προβλήματος και η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που περιμένουν όλοι πώς και πώς θα, πώς θα πρέπει ακριβώς να συμβάλλει στην καλύτερη συνειδητοποίηση της κατάστασης γιατί εκτιμήσεις ε, κινδύνου και ιστοσελίδες ε, για αξιολόγηση του κινδύνου, για εκτίμηση του κινδύνου, ώστε να εντοπιστούν κάποιες συμπεριφορές που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες ή που επιτείνουν τον κίνδυνο, είναι χρήσιμε, χρήσιμες για τους γεωργούς. Γιατί έχουμε αφενός μηχανικούς κινδύνους, αλλά και κινδύνους για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ιδιαίτερα για τα παιδιά, γιατί πολύ συχνά έχουμε πολύ σοβαρά ατυχήματα στις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν επίσης υγειονομικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι στην κυκλοφορία, όπως σας είπα. Έχουμε ένα τεράστιο φάσμα κινδύνων λοιπόν και γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε αυτό το τεράστιο έργο της εναρμόνισης, γιατί έχουμε διάφορες νομοθετικές διατάξεις, γιατί λοιπόν να μην ασχοληθούμε και με τις νομοθετικές διατάξεις που θα διέπουν την υγεία και προστασία των γεωργών. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνας. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Τόμας Λίαμ, πολύ καλά που οργανώσατε την ε, σημερινή εκδήλωση. Θα χρειαστεί να φύγω δυστυχώς προώρα, αλλά είναι πολύ καλή ιδέα και πρέπει να κάνουμε πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Απλώς για να διευκρινίσω ένα-δύο ζητήματα. Υπάρχει διαφορά ως προς την στάση σε σχέση με την ασφάλεια μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εκμετάλλευση. Μετά μας είπατε ότι η Ζηλανδία έχει χαμηλότερο επίπεδο θανάτων στην ε, γεωργική δραστηριότητα, στην ε, γεωργική εκμετάλλευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εάν άκουσα καλά, εάν κατάλαβα καλά, θα μου εξηγήσετε γιατί. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μια χώρα η οποία έχει μεγάλη ένταση γεωργίας και ίσως είναι ενδιαφέρον αν πράγματα έχει χαμηλότερα ποσοστά από εμά να δούμε γιατί. Σε σχέση με τις χημικές ουσίες η νομοθεσία μας εφόσον ε, εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη, φανταζομαι ότι θα έπρεπε να έχει ε, πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να εξετάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Η Ιρλανδία, τουλάχιστον δική μου πατρίδα, φροντίζει ιδιαίτερα να ε, καταρτίζει για την χρήση των μηχανημάτων, των ουσιών κτλ., των χημικών ουσιών και γι' αυτό έχει και χαμηλά ποσοστά. Μήπως πρέπει να επεκταθεί αυτό το μέτρο και αλλού η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση έχει τεράστια σημασία. Πρέπει δηλαδή ο Γεωργός να καλοσκέφεται πριν χρησιμοποιήσει κάτι το επικίνδυνο. Εγώ πολύ συχνά λέω στο Γεωργό δεν, δεν εκτιμάτε αρκετά την δική σας τη ζωή και την υγεία. Αυτό πρέπει να προσέξετε πιο πολύ. Πώς λοιπόν μπορούμε να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση. Και επίσης εάν υπάρχουν πρότυπα που μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως μια γεωργική εκμετάλλευση πρότυπη, η Φερρυπίν ε, γαλακτοκομείο που μπορεί να λειτουργεί με βάση τους κανόνες της υγείας και ασφάλειας και να αποτελέσει παράδειγμα, υπόδειγμα για τους υπόλοιπους. Και... Μια και συχνά μιλάμε για οικογένειες, για παιδιά που χάνουν τη ζωή τους ε, για την ανάγκη και φροντίδα όσων έχουν τραυματιστεί μόνιμα και την ανάγκη να προαγάγουμε την υγεία και ευαισθητοποίηση μέσω της οικογένειας περισσότερο και όχι μέσω στόχο των εργαζόμενων ή των γεωργών μόνο. Εδώ θα ήθελα λοιπόν τις ιδέες σας. Και επίσης, Πρόεδρε, μπορούμε να έχουμε δύο εκθέσεις. Η Επιτροπή Γεωργίας με τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα μελήματα σχετικά με την εργασία του εργαζομένου. Ε, μπορεί να δώσει μια οπτική και από την άλλη η Επιτροπή Γεωργίας με τα δικά της τα θέματα, την νομοθεσία και τον τρόπο εργασίας, ειδικά στη γεωργική εκμετάλλευση του Γεωργού. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τη γνώμη σας. Χίλιες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί από ό,τι ακούμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να δώσουμε λύσεις. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι θα συζητήσουμε διάφορα θέματα αρμοδιοτήτων των επιτροπών. Δεν είναι πάντα εύκολο. Η κυρία Σάιρουκ τώρα. Από τους Σοσιαλδημοκράτε για την κοινωνική πολιτική πάντα αρμόδια. Γιώτα, έχει το λόγο. Ναι, πρόεδρε, πολύ στομα. Ευχαριστώ όλου του ομιλητές. Δείξατε, νομίζω, αφενός ότι η γεωργία είναι ένα θέμα που σπάνια συζητούμε, ίσως δική μας ε, ε, Επιτροπή με τη διάσταση της υγείας και της ασφάλειας, αλλά από την άλλη σημειώνεται πόσο σημαντικό είναι και η Γεωργική Επιτροπή να συζητεί πάντα, αλλά και η Επιτροπή Απασχόλησης. Πρέπει μονίμως να μας απασχολεί το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στη Γεωργία. Μας έχουν ε, απασχολήσει θέματα υγείας και ασφάλειας κατά περίπτωση όταν είχαμε να κάνουμε εποχιακούς εργαζομένους ή με ε, μετανάστες εργαζομένους όπου προσπαθούσαμε να ενισχύσουμε τη θέση των εργαζομένων και είχαμε καταφέρει μάλιστα να προωθήσουμε έναν ε, ε, ουσιαστικό τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι και το γεγονός ότι είναι πολύ διαφορετικές οι εκμεταλλεύσεις γιατί εγώ, ε, παραδείγματι, από μια περιοχή της ε, Γερμανίας που γνωρίζει μικρές και μεσαίες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, γνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ε, ότι μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερες σε άλλες περιοχές με τελείως διαφορετικά και δικά τους προβλήματα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε το ζήτημα της ε, στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι, ε, και ίσως με ιδέες για προστασία, συστάσεις, ε, να μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την υπηρεσία που ασχολείται με το θέμα αυτό, την αποκεντρωμένη υπηρεσία. Εμείς επισκεφθήκαμε τον Πιλμπάο πρόσφατα ως αντιπροσωπεία και ίσως θα ήταν καλό και σε ένα άλλο σημείο της ημερήσιας διάταξης να κοιτάξουμε, δεν ξέρω προβλέπετε, ε, το θέμα αυτό και την ε, συνέχεια που θα δοθεί στην υπόθεση αυτή. Υπάρχουν ανάγκες, υπάρχει ανάγκη για δράση, το είπαμε αυτό, και υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που καταγράφονται για την υγεία και την ασφάλεια στο μεγάλο αυτό κλάδο, όπως τα λέγαμε, της Ευρώπης. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε κάποιες δραστηριότητες ομοθετικού τύπου Λόγος πολλής έχει γίνει επίσης για βέλτιστες πρακτικές, για υποδειγματικές πρακτικές, για παραδείγματα, καλά παραδείγματα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δώσατε κάποιες συγκεκριμένε ιδέες με λύσεις ε, που ενδεχομένως έχουν εξευρεθεί και θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ε, θέση των γεωργών. Εγώ θα ήθελα να πω και με ενδιαφέρει το εάν, ε, και εσείς ως ειδικοί σε αυτήν την ιδέα, το εάν οι μικρότερε εκμεταλλεύσει αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα από την παρατήρησή σας ως προς την προστασία της υγεία υγείας και της ασφάλειας, του τρόπου εργασίας δηλαδή και πώς, εν πάση περιπτώσει, τους εργαζόμενους στα εκμεταλλεύσεις αυτές μπορούμε να τους προστατεύσουμε καλύτερα. Γιατί και στα φυτοϊγειονομικά, τα ε, χημικά που χρησιμοποιούνται, αλλά και τα λοιπάσματα χρειάζεται να κοιτάξουμε με πολύ πιο μεγάλη προσοχή τι θα εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριο Μπένι από του Φιλελευθέρου, πάντα δυναμικό και αποφασιστικό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Να αναφέρω την προσωπική μου εμπειρία, αν μου το επιτρέπετε. Η πρώτη εμπειρία που είχα με τους κινδύνους ενός αγροκτήματος είναι όταν ήμουνα τριών ετών έσπρωχνα ένα καροτσάκι και ο πατέρας μου πέρασε δίπλα με ένα τρακτέρ και ουσιαστικά το, το έριξε, με έσπρωξε με αυτό. Και έκτοτε πρέπει να σας πω ότι σε ένα τέτοιο τελικά περιβάλλον μεγάλωσα, σε ηλικία 12 ετών, α, ράντιζα κάποια φυτά χωρίς να έχω όμως την απαραίτητη προστασία. Σταμάτησα βέβαια να χρησιμοποιώ τους φωσφάτες αυτούς όταν ανέλαβα εγώ την γεωργική παραγωγή γιατί ε, συνειδητοποίησα ότι ε, δεν ήταν καλά τελικά αυτά οι ουσίες αυτές για την υγεία μου, γιατί με έπιανε φαγούρα λίγες ε, ώρες αφού τα είχα χρησιμοποιήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καλό το ότι δεν χρησιμοποιούμε πλέον κάποιες από τις πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούσαμε στη Γεωργία στο παρελθόν. Τώρα τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε κάποιες πολύ αυστηρές κατευθυντήρες γραμμές όσον αφορά την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών. Και νομίζω ότι καταβάλαμε πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί η χρήση των χημικών αυτών ουσιών. Και μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες ενημέρωσα έναν εργαζόμενό μου για, τις ασφαλείς, για την ασφαλή χρήση των ουσιών αυτών και του ζήτησε επίση να κάνει και του απαραίτητου ελέγχου. Το πρόβλημα όμω είναι ότι συχνά οι άνθρωποι που εργάζονται μόνοι του, οι αυτοαπασχολούμενοι, δεν προσέχουν τόσο πολύ. Πάρα πολύ σκέφτονται ότι μόνος μου θα χρησιμοποιήσω το αλυσοπρίο μου, μόνος μου θα χρησιμοποιήσω τις χι χημικές ουσίες και δεν υπάρχουν όμω τότε οι οι έλεγχοι. Το βασικό ζήτημα πάντως που θέλω να θίξω είναι ότι Αυτό το οποίο είπατε και εσείς, η εκστρατεία που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν ένας από τους γεωργούς αυτούς που πήγαν και παρακολούθησαν μία από τις μερίδες αυτές. Και πρέπει να σας πω ότι ε, παραπονιόμασταν τότε ότι μας είχατε αποστείλει μια επιστολή και μας είχατε πει ότι αν δεν παρακολουθούσαμε το μάθημα αυτό, τότε θα μας γινόταν μια επιτόπου επιθεώρηση. Και Όλοι οι γεωργοί που γνωρίζω ουσιαστικά παραπονιό, παραπονιόντουσαν όλοι και γκρίνιαζαν. Ήρθαμε λοιπόν στο μέρος αυτό που είχε προβλεφθεί για την ημερίδα αυτή και μπορώ να σας πω ότι τελικά όλοι κάτι κερδίσαμε από τις πάρα πολύ καλές αυτές παρουσιάσεις που μας γίνανε για τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, συγκεκριμένα στη γεωργική εκμετάλλευση. Θεωρώ ότι τέτοια παραδείγματα πρέπει να γίνονται πρακτικοί σε πάρα πολλές χώρες. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό είχα πάλι ένα ατύχημα στην δική μου τη γεωργική εκμετάλλευση. Την τελευταία στιγμή κατάφερα να αποφύγω το ατύχημα, είχε να κάνει με τη χρησιμοποίηση μιας σκάλας. Αλλά ξέρετε ότι αντίστοιχα ατυχήματα μπορούν να συμβούν και με άλλο γεωργικό εξοπλισμό. Όσον αφορά τη Νέα Ζηλανδία, νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η γεωργική τους παραγωγή διαφέρει τελικά από την δική μας γεωργική παραγωγή. Ουσιαστικά δεν αναγκάζουν να χρησιμοποιήσουν τόσο συχνά κάποια από τα γεωργικά μηχανήματα τα οποία εμείς εκτενώς χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Τα εξκαφικά, για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούνται τόσο εντατικά στη Νέα Ζηλανδία όσο χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ πάντω ότι θα ήταν πάρα πολύ θετικό όλε αυτέ οι πρακτικέ ενημέρωση να αρχίσουν να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και τώρα θα μα δώσουν ένα καλό παράδειγμα και υπόδειγμα πλήρου πειθαρχία οι εμπειρογνώμονέ μα. Τέσσερα λεπτά ο καθένα είναι δυνατόν, παρακαλώ. Α ξεκινήσουμε από τι κυρίε. Ladies first. Η κυρία Πόντνιτσε, έχετε το λόγο. Τρία, λεπτά. Τρία λεπτά. Και αν μου επιτρέψετε θα σας κάνω νέο ημό όταν τελειώσω το τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχήν, αν υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Συνήθως ε, οι άντρες είναι πιο ριψοκίνδυνη αυτή η φαλοκρατική νοοτροπία δεν έχουν επίγνωση του κινδύνου. Και αυτό είναι κοινό περισσότερο στον κατασκευαστικό κλάδο και στη Γεωργία. Τώρα, δεν μπορούμε να φτάσουμε όπως σας είπα στον κάθε γεωργό, στην κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Ε, συνεργαζόμαστε με κάποιους μεσάζοντες, ε, για παράδειγμα με κάποιες οργανώσεις που έχουν μέλη γεωργούς σε όλες τις χώρες. Επίσης, έχουμε και τα εθνικά μας ε, σημεία επαφής και εκεί έχουν ε, τριμερή δίκτυα και απασχολούν και εμπειρογνώμονες. Έτσι μπορούμε να διαδώσουμε τις καλές πρακτικές σε όσο το δυνατόν περισσότερους γεωργούς. Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν οι γεωργοί ότι η υγεία τους είναι πολύτιμο αγαθό και αν τους συμβεί κάτι, οι συνέπειες ε, ε, θα επεκταθούν και στην οικογένειά τους και στις επιχειρήσεις τους. Ευχαριστώ κύριο Φρανσουά. Έχετε την ε, ευτυχία και την τύχη να μας μιλήσετε για τρία ακόμη λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ως προς πρακτικές. Ε, όλοι μιλάνε για βέλτιστες πρακτικές. Ωραία. Ναι. Ας μιλήσουμε για αυτές. Αλλά για τα χημικά προϊόντα νομίζω ότι πρέπει απλώς να επικρατήσει κοινή λογική. Όταν είναι επικίνδυνο προϊόν πρέπει να αποσύρεται γιατί ο Γιώργος δεν μπορεί πάντα να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές που ενδεχομένω προβλέπονται. Εάν δούμε λοιπόν τις χώρες που έχουν τη λεγόμενη πλήρη, το πλήρη εξοπλισμό προστασίας, όπως ονομάζεται στη Γαλλία, ολόκληρη τη φόρμα δηλαδή, δεν ε, εφαρμόζεται. Στην ε, δε Γαλλία πρέπει να πω ότι έχει δύο ημέρες υποχρεωτικής κατάρτισης ο, Γερμανός, ο Γάλλος Γιώργος, όχι μισή, ε, για να πιστοποιηθεί. Αλλά πάνω απ' όλα απαραίτητο είναι να επικρατεί η κοινωνική. Από την άλλη βέβαια μετά υπάρχουν οι διάφορες πρακτικές στον χώρο εργασίας και όλοι οι λοιποί που παρεμβαίνουν. Ο... Ε, πέραν του Γεωργού, ο ε, κλαδευτής που θα έρθει για να κλαδέψει το αμπέλι, επί παραδείγματι το κλίμα, ε, εξαρτάται από το τι είδους χημικά έχει χρησιμοποιήσει πριν από αυτόν ο απελουργός Και ούτω καθεξής. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται τώρα για διαταράκτες ενδοκρινικούς, πρόκειται για πολύ ε, τοξικά προϊόντα. Αλλά πάνω απ' όλα, όπω είπα, πρέπει, γιατί οτιδήποτε και να εφαρμόζεται, ε, οτιδήποτε και να ισχύει δεν απαραίτητο να εφαρμόζεται όπω πρέπει στην πράξη, πρέπει να επικρατεί η κοινή λογική. Ρωτήσατε για τι γυναίκε. Ναι, οι γυναίκε είναι πιο προσεκτικέ. Και οι γυναίκε πολύ συχνά είναι αυτέ οι οποίε καταγγέλουν τα όσα συμβαίνουν στην Υπεθρό. Είναι πολύ θαραλέ, όχι μόνο προστατεύουν τον εαυτό του, αλλά ε, προειδοποιούν και τους συζύγους τους, γιατί πολύ συχνά είναι αυτές οι οποίες διαπιστώνουν το πρόβλημα υγείας από το οποίο πάσχει και ενδεχομένω δεν αναγνωρίζει ο ίδιος ο Γεωργός. Με το θάρρος λοιπόν που επιδεικνύουν πολύ συχνά είναι οι αγρότες οι οποίες ε, ε καταγγέλνουν αυτές τις πρακτικές. Από την άλλη βέβαια θα έλεγα και υπογραμμίζω δεν θα αρκίσει δεν θα αρκέσει, γιατί οτιδήποτε οδηγούς και εγχειρίδια να συγγραφούν οτιδήποτε ενημέρωση να γίνει και στον Γεωργό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από καθέδρα. Στην καθημερινή ζωή μαθαίνει κανείς. Και όπως είπατε υπάρχουν και οι κλιματικές αλλαγές. Δεν έχουμε μόνο το τρακτέρ. Πολύ σωστά ε, υπογραμμίσατε ότι αυτό μπορεί να σημαίνει σε μια γεωργική εκμετάλλευση όπως η δική μου μπορεί, μεγάλη δηλαδή μπορεί να μην ισχύει κάπου αλλού, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλοι ή μικροί γεωργοί, μεγάλες ή μικρές εκμεταλλεύσεις και από εκεί να εξαρτάται ο κίνδυνος. Όχι, είναι η καλή και η κακή ενημέρωση και κατάρτιση. Ίσως είναι οι συνδικαλιστές του, του τομέα της Γεωργίας δεν μιλούσαν με τους ίδιους όρους όπως εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να μιλάμε για το περιβάλλον, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα χημικά προϊόντα δεν επηρεάζουν μόνο το, το περιβάλλον. Αν ο Γεωργός αντιληφθεί ότι ε, μπορεί να προσβάλλει την ίδια του την υγεία με τη χρήση του, τότε ταυτόχρονα και μοίρα θα προστατέψει και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Κύριος Δελγάτο Κομπάς. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά την προστασία των μικρών γιώργων, των μικροκαλλιεργητών. Είναι δύσκολο για ένα μικροκαλλιεργητή να ασχοληθεί με την πρόληψη στην εκμετάλλευσή του, ιδιαίτερα όταν έχει επικίνδυνες δραστηριότητες. Όταν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα, για παράδειγμα. Με βάση την Ισπανική νομοθεσία, για τέτοιου είδου ουσίε κάποιο ανειδίκευτο δεν μπορεί να εκτιμήσει τον κίνδυνο τη χρήση τέτοιων προϊόντων, αν δεν έχει την κατάλληλη επιμόρφωση κατάρτιση. Γι' αυτό οι γεωργοί πρέπει να προσλάβουν κάποιον ε, που να κάνει την εκτίμηση του κινδύνου, κάποιον εξωτερικό σύμβουλο που πρέπει να είναι ειδικευμένο σε θέματα γεωργίας και μάλιστα ελέγχεται η δραστηριότητα τέτοιου συμβούλου ε, για να εξασφαλιστεί η ποιότητά της. Αλλά δεν μπορούν όλοι οι μικροκαλλιεργητές να, προσλάβουν έναν ε, εμπειρογνώμονα. Γι' αυτό και είπα ότι χρήσιμο θα ήταν τέτοιου είδου ε, υπηρεσίες πρόληψης, ε, ειδικέ για τη γεωργία, να παρέχονται στους μικροκαλλιεργητέ με με κάποια οικονομικά κίνητρα γιατί δεν μπορούν οι ίδιοι να πληρώσουν όλο το, τμήμα, το τίμημα. Ένα τμήμα λοιπόν των ε, επιχορηγήσεων τη κοινή γεωργική πολιτική, καλό θα ήταν να αφιερώνεται στην χρηματοδότηση τέτοιων υπηρεσιών πρόληψη για του γεωργού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ε, φυτογενομικά προϊόντα, φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα κτλ. Εμείς ε, κάνουμε μια αξιολόγηση του κινδύνου της έκθεσης σε τέτοια προϊόντα και μάλιστα συνεργαζόμαστε στην κατάρτιση μητρώου τέτοιων προϊόντων, φυτοφαρμάκων δηλαδή, στην Ισπανία. Με βάση μια οδηγία του 91, την 91-414, ε, βλέπουμε ότι οι δραστικές ουσίες των προϊόντων αυτών είναι ίδιες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ένας κοινοτικός κατάλογος για επιτρεπόμενα προϊόντα με επιτρεπόμενη δραστική αξία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν προϊόντα που δεν περιέχουν τις επιτρεπόμενες δραστικές ουσίες. Βέβαια από το 1991 και μετά αναθεωρείται ο κατάλογος και ελάχιστες ουσίες έχουν παραμείνει εκτός της αναθεώρησης. Θα ολοκληρωθεί και για αυτές ε, εντός ολίγου, οπότε οι δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων αυτών θα είναι ίδιες σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης έγινε σημαντική πρόοδος σε νομοθετικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 2009 δημοσιεύτηκε ο νέος κανονισμός για την εμπορευματοποίηση αυτών των προϊόντων και που ε, κατηγορηματικά απαγορεύει οποιοδήποτε προϊόν που μπορεί να είναι μεταλλαξιογόνο, καρκινογόνο και ούτω καθεξής. Αυτό προβλέπει ο νέος κοινοτικό κανονισμός. Σε ό,τι αφορά τη χρήση, πέρυσι ε, τέθησε ισχύ μία οδηγία για τη βιώσιμη χρήση που περιλαμβάνει και το σκέλος της πρόληψης. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα των φυτοφαρμάκων ε, οριοθετείται σωστά και σε κοινοτικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σόμπος. Και τέλος ο κύριος Πάτρικ Γκρίφινγκ. Από την Ιρλανδία. Να ξακούσουμε λοιπόν και έναν Ιρλανδό Γιώργο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλά θέματα. Θα προσπαθήσω να τα καλύψω όλα. Το προσδόκιμο ζωής είναι μειωμένα όντω για του γεωργού. σημαντικά, δηλαδή πεθαίνουν νωρίτερα οι γεωργοί, πολύ νωρίτερα από οποιονδήποτε άλλο επάγγελμα, είτε από καρδιακιακά, είτε από καρκίνο, είτε ακόμη και από ε, αυτοκτονίες που είναι πιο συχνά στο γεωργικό τομέα, πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει ερωτηματικά. Όντως οι γυναίκες αναλαμβάνουν λιγότερους κινδύνους θα συμπληρώσω όμως ότι εν γέννη οι γυναίκες δεν ε, συμμετέχουν στις πιο επικίνδυνες ε, γεωργικές εργασίες όπως το να χειρίζονται είτε μεγάλα ζώα είτε γεωργικά, βαριά γεωργικά μηχανήματα. Αλλά πολύ συχνά έχω πει ότι αν προέβαιναν σε αλλαγή φίλου γεωργή μπορεί να λύναμε πολλά προβλήματα αυτό ως αστείο. Την ε, τη Νέα Ζηλανδία την παρακολουθούμε και με πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έχει αντίστοιχες με τις ε, Ιρλανδίας γεωργικές δραστηριότητες. Έχουν όμως ε, πάνω απ' όλα κτηνοτροφία προφάτου που σχετίζεται παρουσιάζει χαμηλότερε στατιστικέ θανάτων από αυτή τη ε, αγελαδοτροφία, που είναι το χαρακτηριστικό τη Ιρλανδία. Είναι διαφορετικά τα μηχανήματα και μικρότερη η συχνότητα χρήση βαρέων μηχανημάτων στην Ζηλανδία, στην Νέα Ζηλανδία. Πάντως θα παρακολουθούμε, όπω σα είπα, και αν υπάρχει τρόπο, και βρούμε ε, αντιστοιχίε ή λύσει που θα ήταν χρήσιμε θα τι αξιοποιούσαμε. Οι γεωργοί που λέτε ότι δεν, ε, δεν προσέχουν τη ζωή του. Δεν τιμάνε την ίδια του τη ζωή. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό και στην κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ο Ευρωπαίος πολίτης τιμά τον Γεωργό. Εάν η ίδια η κοινωνία δεν τιμά τον Γεωργό, πώς είναι δυνατόν ο Γεωργός να τιμά τον εαυτό του. Όλοι περιμένουμε είτε στη στο κηλικείο είτε στο σούπερ μάρκετ ε, είτε στο εστιατόριο να βρούμε έτοιμο το φαγητό, αλλά το θέλουμε και φθηνό Δεν είμαστε τεθειμένοι να το πληρώσουμε ακριβά. Πράγμα το οποίο σημαίνει μετακύληση των προβλημάτων στο Γιώργο. Πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να πληρώνουμε πιο με υψηλό τίμημα για την τροφή μας, για να πληρώνεται καλύτερο ο Γεωργόρος να είναι παραγωγικός, χωρίς να διατρέχει κινδύνους. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Επίσης, κάνουμε ε, με υποδειγματικές εκμεταλλεύσεις την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των γεωργών. Πολλές φορές το έχουμε κάνει αυτό. Υπάρχουν όλες, πολλά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και ε, λύσεις που έχουν αποδώσει και στην ε, Δανία, επί παραδείγμα στη Δυτική Ιωτλάνδη. μπορούμε να δούμε αντίστοιχα παραδείγματα από ο Ηνωμένο Βασίλειο, που όμως ήταν πολύ δαπανηρά με εκμεταλλεύσεις που κόστησαν και 10.000 ευρώ την ημέρα ως κόστος λειτουργίας. Πήγα εγώ, τα επισκέφθηκα, αλλά ίσως θα πρέπει να παρεύει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να στηρίξει τις προσπάθειες. Πάντως, η όλη προσέγγιση είναι ότι χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής. Τα κράτη-μέλη έχουν προσφέρει την καθοδήγησή τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης τώρα, αλλά οι θάνατοι και τα σοβαρότατα ατυχήματα στις ιερουργικές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν πάψει. Ε, δεν αρκεί, δεν δίνεται λύση με τη δημοσίευση εγχειριδίων και οδηγών. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και για την ε, αναστροφή των δημογραφικών τάσεων στον χώρο της γεωργίας, γιατί είναι πολύ ηλικιωμένη η γέννη γεωργία στην Ευρώπη. Χρειάζεται καλύτερη κατάρτιση, αλλαγή πολιτικής ώστε να, αξιο... να αξιολογείται ο κίνδυνος στον χώρο της γεωργίας και μια νέα στρατηγική για την υγεία και την ε, ασφάλεια στον χώρο εργασίας, όταν αυτός ο χώρο εργασία είναι η γεωργία. Άρα λοιπόν πολιτική αλλαγή, αλλαγή πολιτικής και όχι διαρκής ε, εκδόσεις ε, ε, αλλεπάλληλες εκδόσεις οδηγών και εγχειριδίων. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής στη Γεωργία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και για τα καταληκτικά σχόλια. με εσύ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι από τα όσα ακούσαμε σήμερα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή η συζήτηση αυτή εφόσον συζητούμε την μεγαρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, ακόμα και στα πλαίσια της πρόοδου που επετεύχθη χθε από το Συμβούλιο, χθε το βράδυ. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβλεφθούν, αν μη τι άλλο, κάποιες διατάξεις στα πλαίσια της νέας αυτής κοινή γεωργικής πολιτικής για να αυξηθούν τα πρότυπα ασφάλεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Είναι ζωτική σημασία να γίνει κάτι τέτοιο ευαισθητοποίηση, καλύτερη ενημέρωση, βέλτιστε πρακτικέ. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα ζητήματα αυτά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σαφώ ευρωπαϊκή διάσταση σε όλα αυτά, παράλληλα με την εθνική δραστηριότητα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Μου κάνει εντύπωση που βλέπω ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν καθόλου στατιστικά δεδομένα. Αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πίεση και για αυτό το ζήτημα. Τώρα, κάποιες ε, βέλτιστες πρακτικές, η αύξηση των ερευνών, το να χρησιμοποιούμε όλο και πιο ασφαλή μηχανήματα, καλύτερες πρακτικές επιτόπου. Όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν πάρα πολύ καλά, αρκεί να μπορούν να αλλοιοποιηθούν βέβαια οι πρακτικές αυτές. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι στην προσπάθειά μας να αυξήσουμε την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία μπορούμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω άχθος και περιορισμού στη γεωργική δραστηριότητα. Το τελευταίο το οποίο θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να βαρύνουμε ακόμα περισσότερο τον ήδη βαρύ κατάλογο πολλαπλής συμμόρφωσης που ισχύει για τους γεωργούς. και ότι δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπω στα ύδατα, τα θέλετε, της δικής σας Επιτροπής Απασχόλησης, πιστεύω ότι εμείς, τουλάχιστον στην Επιτροπή Γεωργίας, μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα πολύ ζωτικό ρόλο. Το είδαμε αυτό σήμερα. Δηλαδή να διευκολύνουμε τη μελλοντική συζήτηση για τα ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν σήμερα. Να καταλήξω τέλος ευχαριστώντας τους ε, ανθρώπους που ήρθαν εδώ πέρα σήμερα για να μας ενημερώσουν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και το πιο σημαντικό είναι η συζήτηση αυτή να, μας, να μην σταματήσει εδώ σήμερα. Να δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση αυτή και να καταφέρουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Ιδίω αυτή τη χρονική στιγμή που συζητάμε και την πραγματευόμαστε τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτική. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχουμε νομίζω μια πολύ καλή ε, εικόνα εξασφαλίσει. Βλέπουμε από τις δύο επιτροπές ότι είναι το θέμα το οποίο είναι πολύ επίκαιρο, μας ενδιαφέρει πολύ και πρέπει νομίζω να ομολογήσουμε ότι και οι πολιτικοί είναι σε θέση να ακούνε, να προσέχουν, να τίνουν νους δεν αποστρέφονται τον ομιλητή του. θέλουν να ακούνε συγκεκριμένε προτάσεις και αυτά μπορέσαμε όλα να τα κάνουμε σήμερα. Ενημέρωση, κατάρτιση, εκπαίδευση, πιστοποίηση εκπαίδευσης, δυνατότητα εντοπισμού των κυρίων πηγών κινδύνου, ε, αποθηκευτική χώρη, εργοτάξια, ηλεκτρομαγνητικά πεδία που ανέφερε και η Ελίζαμπετ και που έχουμε για τον τριμερή διάλογο μπροστά μας, ένα πολύ δύσκολο θέμα. Τομεί λοιπόν που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και δεν πρέπει να λησμονούμε και το άλλο θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε, που είναι ο χρόνος εργασίας, οι ώρες εργασίας, που πρέπει Πολλέ φορές νομολογήσουμε ότι διαμορφώνονται έτσι ώστε πλέον υπάρχουν απορρέων κίνδυνοι μόνο και μόνο από τι ώρε εργασία. Επίσης, η νομική υποστήριξη. Πώ μπορεί δηλαδή κανεί να γνωρίζει, να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του και να μην χρειάζεται να περιμένουμε κάθε φορά μια μη κυβερνητική οργάνωση να τον, να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν προβλήματα υπάρχουν και στα φυτοϊγειονομικά αλλά και σε άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σημαντικά προβλήματα και πρέπει να τα προσέξουμε. Με μια από τις παρατηρήσεις λοιπόν που θεωρώ πολύ σημαντική θα ήθελα να ολοκληρώσω σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω τη φράση που ακούστηκε ότι πρέπει να στραφούμε προς τον καταναλωτή και να μεριμνήσουμε για χάρη του καταναλωτή να έχουμε όχι μεγάλες ποσότητες, όχι πάντα ένα γεμάτο τραπέζι, ε, ίσως πιο λιτό τραπέζι, αλλά πάντως ποιοτικό τραπέζι, ποιοτικά προϊόντα, καλά προϊόντα και σε αυτό θα πρέπει να στραφεί η παραγωγή της γεωργίας. Και γι' αυτό πρέπει και ο γεωργός να εισπράττει, να αμείβεται με καλά ποσά, με ικανοποιητική αμοιβή, ώστε να μπορεί να διατηρεί αυτή την ποιοτική δραστηριότητα. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερως. Είχαμε, νομίζω και οι δύο επιτροπές συμφωνούμε, εξαιρετικούς ε, ομιλητές και ειδικού ε, δεν είναι εύκολο πάντα να γίνεται μια κοινή συνεδρίαση επιτροπών με ακροάσει, αλλά νομίζω τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα διακόψω για μερικά λεπτά προκειμένου να συνεχίσουμε μετά με την ε, υπόλοιπη μερίσια διάταξη και πάλι ευχαριστώ θερμά του εδώ παρισταμένους ομιλητέ και συναδέλφου. Σας ευχαριστώ λοιπόν κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ οι διμερείς συνομιλίες εκτός εθούσης, γιατί εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Δύο λεπτά παρακαλώ υπομονή Τζιν. So, Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Υπάρχουν και εκτός αιθούσης ε, καταπληκτικές γωνιές για να συνεχίσετε τις συνομιλίες σας. Στο σημείο 13, συνέπειες της κρίσεως, πρόσβαση στην φροντίδα για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Τζιν Λάμπερτ. Επιπτώσει κρίσεων αφορά την προσβάση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη. Η Τζιν λοιπόν ε, δεν μιλάει γερμανικά, αλλά ξέρω ότι τα καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και πάντω εννοούμαστε πάρα πολύ ωραία με τα αγγλικά τη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώ η γνώση μου των γερμανικών περιορίζεται σε παραγγελίε ποτών. Θα εξετάσουμε σήμερα τις τροπολογίες της έκθεσης μου που αφορά την πρόσβεση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη. Θα διαπιστώσετε ότι έχουν κατατεθεί 157 τροπολογίες, πληθώρα τροπολογιών. Μερικές βέβαια είναι δικές μου. Πάντως, εν γέννη, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τροπολογιών είναι πολύ επικοδομητική Έχουμε κάποια νέα στοιχεία για την ε, γεωργική διάσταση, για την συμπερίληψη της υπαίθρου, την πρόσβαση, τη δυσκολία πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ούτω καθεξής. Δεν μπορούσαμε να περιορίσουμε την έκθεση μόνο στην υγειονομική περίθαλψη, ε, γιατί είναι αρμόδια, είναι αρμόδια και Επιτροπή Περιβάλλοντος γι' αυτό. Μιλήσαμε φυσικά για τις αναπηρίες, την υγειονομική περιθέλψη, τους ηλικιωμένου και τα παιδιά, που είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες. Ή ε, τα παιδιά που για κάποιους λόγους δεν ε, βρίσκονται με την οικογένειά τους. Μερικές τροπολογίες προτείνουν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή έκθεση και συμπερίληψη και νέων πτυχών για παράδειγμα, αναφέρονται στην ενεργογύρανση ή κάποιες μεταρρυθμίσεις του, των συστημάτων υγείας. Ε, τροπολογία 63 του κ. Σάμπρνοχ, για παράδειγμα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε αν θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο την εμβέλεια της έκθεσης. Αν η πλειοψηφία το κρίνει απαραίτητο και σκόπιμο, δεν θα εκφράσω εγώ αντίρρηση. Σε ό,τι αφορά τις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Για παράδειγμα, αυτούς που ασχολούνται με τη φροντίδα ε, και κυρίως όσους αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας ή σε οικογενειακό περιβάλλον. Παράγραφος 12 παράγραφος 21 από αυτών των θεμάτων. Θα προσπαθήσουμε στις παραγράφους αυτές να καταλήξουμε συμβαστικές προτάσεις για τις εργασιακές συνθήκες στον τομέα. Επίσης το δυναμικό σε θέση απασχόλησης, κάτι που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικά της έγγραφα. Ένα τρίτο θέμα η υποστήριξη ε, των ε, μελών της οικογένειας ε, που ασχολούνται με την φροντίδα και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την παροχή τέτοια φροντίδας. Επίσης, μια οδηγία που αφορά την άδεια για αυτούς που παρέχουν φροντίδα. Και τα αποτελέσματα, οι συνέπειες τις υποχρέωσης παραγωγής φροντίδας για τις γυναίκες και πώς αποποιεί αυτό την κατάστασή τους σε σχέση με άλλες αμοιβόμενε εργασίες. Μερικές τροπολογίες πραγματεύονται για το πώς εξετάζουμε το, τον αντίκτυπο κάποιων αλλαγών που προέκυψαν από την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας των μεταρρυθμίσεων που θεσπίζουν τα κράτη-μέλη και πώς μπορούμε να τις αξιολογήσουμε στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα στοιχεία να τα συνδυάσουμε για να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Άλλες τροπολογίες ε, μιλούν για την ε, χρήση των κοινοτικών κονδυλίων ε, για κατάρτιση, σύνδρομη και ούτω καθεξής. Άλλες τροπολογίες μιλούν για το ειδικό ταμείο για του απόρου. Και εδώ με ενδιαφέρει το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτό το ταμείο έχει κάποια σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα. Γιατί ναι, μεν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, είναι σχετικό με το θέμα που μας ενδιαφέρει, αλλά δεν ξέρω αν το Ταμείο Απόρων είναι το κατάλληλο το ταμείο για να το συνδέσουμε με το θέμα αυτό της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη. Και έχουμε και μεμονωμένα ζητήματα σε κάποιες τροπολογίες, αλλά αυτά θα τα δω διμερός με τους συντάκτες τροπολογιών, για να μην κουράζω την Επιτροπή με λεπτομέρειες. Πάντως, επαναλαμβάνω, οι περισσότερες τροπολογίες είναι πολύ επικοδομητικές είτε εμπλουτίζουν κάποιους παραγράφους, είτε προσθέτουν κάποιους παραγράφους και πιστεύω ότι μετά την περάτωση της διαδικασίας της εξέτασης και της ε, σύνταξης συμβαστικών τροπολογιών θα έχουμε ένα πολύ αίσιο αποτέλεσμα. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας αποφάσισε ότι θα εκπονήσει και αυτή η γνωμοδότηση και γι' αυτό συχάσατε την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Ίσως θα έχετε την ευκαιρία στα πλαίσιο μιας ε, γνωμοδότησης επιτροπή Γυναικών, για παράδειγμα, να καταθέσετε τι τροπολογίες, αλλά παρακαλώ ε, να είστε αρκετά συγκρατημένοι. καλό είναι να μην υποβληθούν πολλέ τροπολογίες. Και είμαι στη διάθεσή σας για να εξετάσουμε το θέμα, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Γιούτα Στάινμπρουκ. κυρία Σίπρα, τη είναι στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών σε μια πολύ σημαντική συζήτηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και γι' αυτό με παρακάλεσε να ε, παρουσιάσω εγώ τις δικές της ε, τοποθετήσεις. Η ΣΥΠΛΙΣ λοιπόν, αλλά και γενικώ από πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τη φροντίδα είναι θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί να περικοπεί, να περιοριστεί ούτε σε περίοδο κρίσεως. Αυτό θα πρέπει να προσφέρεται σε, όλους τους, σε όλες τις ομάδες ε, με τους ίδιους όρους και την ίδια ε, πλοχεριά. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις, ε, τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για την πρόσβαση στην φροντίδα, φερρυπίν, τέλος για παροχή ε, για είσοδο στα νοσοκομεία, παροχή για την φαρμακευτική ε, περίθαλψη στα νοσοκομεία στην Ελλάδα, άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, πολιτική των περικοπών που γίνονται και που μπορεί να έχουν, των περικοπών που γίνονται και μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Ακόμη μέχρι τώρα όχι σαφείς. Οι προτάσεις της Jean Lambert είναι εξαιρετική βάση ε, για συζήτηση. Οι τροπολογίε μας ε, ακολουθούν λίγο πολύ την ίδια κατεύθυνση με την εισηγήτρια και απλώς ενισχύουν το κείμενό τη. κυρία Ζήπερτς είναι πεπισμένη ότι οι τροπολογίε της θα αποτελέσουν μια ευρύτατη βάση συμβιβασμού. Ε, και αναμένει κυρία Ζήπερτ την περαιτέρω συνεργασία στο σημαντικό αυτό θέμα, συνεργασία τόσο με την εισηγήτρια όσο και με τους λοιπούς και όλους τους Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριο Μπέκερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια. Ξεκάθαρα και πρώτα απ' όλα για τον τρόπο της συνεργασίας που μας προσέφερε. το φάσμα θεμάτων ε, που μας απασχόλησαν, ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να εστιαστούμε, να επικεντρωθούμε σε εκείνα τα θέματα που είναι τα πιο σημαντικά, τον ορισμό του ποιο είναι αυτός που χρειάζεται φροντίδα ή προστασία και την αναγνώρισή του. Βέβαια και η φροντίδα και η ε, περίθαλψη έχουν πολύ μεγάλη σημασία εν γέννη για τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτε μας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ ωστόσο στο γεγονός ότι αυτή η έκθεση προσφέρει μία πολύ πλήρη και περίπλοκη ε, έκθεση παρουσίαση δηλαδή, του θέματος και μπορεί να αποτελέσει έναυσμα σοβαρό και σημαντικό για την προαγωγή αυτών των ε, μέτρων, γιατί είναι επιτέλεση του έργου μας κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό ακόμη και δύο ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Μερικά ζητήματα θα χρειαστεί να διευκρινιστούν ασφαλώς, αλλά ουσιαστικά συμφωνούμε με την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Αν όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Δεν χρειάζεται, επομένως ξαναδίνουν το λόγο στην εισηγήτρια. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις επικοδομητικές παρατηρήσεις τους. Όντως, οι περισσότερες τροπολογίες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σημεία σύγκρουση ή αποκλήσει, ενδεχομένω να δίνουμε αλλού την έμφαση σε κάποια σημεία. Όσον αφορά, για παράδειγμα, το θέμα του στίγματος, αν στιγματοποιούνται κάποιες κατηγορίες. Θα προσπαθήσω πάντως να σας προτείνω κάποιες ιδέες για να καταλήξουμε μετά το Πάσχα, μετά το διάλειμμα για το Πάσχα, σε έναν συμβιβασμό. Φαντάζομαι ότι αρκετά αργά στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή, επομένως έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Βάσει λοιπόν αυτών θα συζητήσουμε στις 29 Μαΐου τις συμβαστικές τροπολογίες, άρα η συγγήτρια έχει αρκετό χρόνο μπροστά της για να εκπονήσει αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Όρη, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Ντόιτς, ο οποίος είναι ο εισηγητής μας για την γνωμοδότηση αυτή όσον αφορά την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά τη Ένωση, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τι διαδικασίε που στηρίζουν τι διαπραγματεύσει σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τη Ένωση στι αγορέ δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών. Πρόκειται για γνωμοδότηση την οποία εμεί υποβάλλουμε προ την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, όπου ο Ντανιέλ Κάσπαρη είναι ο εισηγητή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Βρισκόμαστε στη φάση εξέτασης του σχεδίου γνωμοδότησης, για το οποίο ο εισηγητής έχει προτείνει έξι τροπολογίες. Κύριε Όρη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όντως χρειάστηκε να επιστρέψει στην Ουγγαρία ο κύριος Ντόιτς, γι' αυτό μου ζήτησε να παρουσιάσω στη δική του τη θέση την γνωμοδότηση την οποία συνέταξε μου άφησε κάποιες σημειώσεις προκειμένου να μπορώ να κάνω μια παρουσίαση. Καταρχάς θα ήθελε να τονίσει πόσο σημαντικές είναι οι δημόσιες συμβάσεις οι οποίες καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο χώρο και όλο και σημαντικότερη θέση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και γενικότερα στον τρίτο κόσμο. Αναφερόμαστε σε ένα 16% πλέον, αυτό είναι το μέρισμα των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση, 11% στις ΗΠΑ, 19% στην Ιαπωνία και στην Κίνα αντιστοιχεί το ποσοστό αυτό στο 15%. Αρκεί βέβαια να έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία είναι αξιόπιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν τομέα πολύ σημαντικό. Από την άλλη βλέπουμε ότι ε, οι δημόσιες συμβάσεις ε, υπάρχονται σε εντελώ διαφορετικούς κανονισμούς από τη μία χώρα στην άλλη. Πάντως αντιστοιχούν σε πολύ σημαντικά ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, και ευρωπαϊκές χώρες αλλά και μη ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να προκυρήσουν διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε για ένα ποσό 550 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ιαπωνία έχει ένα ποσοστό ανοίγματο 28%, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν τελικά μεγάλες αποκλίσεις από τη μία περιφέρεια στην άλλη, από τη μία χώρα στην άλλη. Ο κύριος Ντόιτς εξέτασε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τα παρέτα μέσα προκειμένου να επιτρέπει σε τρίτε χώρε, σε εταίρου Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν πρόσβαση στην ιστορική αγορά τη Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Και μάλιστα υφίσταται μία συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε, προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει όσον αφορά τι ε, εμπορικέ συμφωνίε να μπορούν δηλαδή να περιέχουν και τη διάσταση των δημοσίων συμβάσεων. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία, εφόσον συναυθεί, θα είναι η σημαντικότερη εμπορική συμφωνία παγκοσμίω. Καταλαβαίνετε ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πρέπει επίση να πούμε ότι χρειαζόμαστε και μία διεθνή πλέον ρύθμιση Σήμερα βλέπουμε ότι ένα 25% δραστηριοτήτων των Ευρωπαίων, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συνδέονται με δημόσιες συμβάσεις. 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αντιστοιχούν σε αυτές τις συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ταμας θεωρεί ότι πρέπει να τονίσουμε την κοινωνική σημασία των δημοσίων συμβάσεων. Η κοινωνική πτυχή θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας και θα πρέπει να τονίσουμε όλα αυτά τα κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική αυτή διάσταση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υφίστανται οι καλύτερε δυνατέ συνθήκε προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσει εργασία και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αύξηση και διατήρηση των θέσεων εργασία. Και θα πρέπει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα κατάλληλα μέσα που θα τη επιτρέψουν να καταλήξει σε ισορροπημένε λύσει στι τρίτε χώρε αλλά και στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να συμμορφωθούμε με όλου του υφιστάμενου κανόνε προστασία τη απασχόληση, να συμμορφωθούμε με όλου του υγειονομικού κανόνε και με τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και θα πρέπει να συμμορφωθούμε και με όλου τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες που υφίστανται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που νομοθετούμε στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Στα σημεία αυτά επιμένει άλλωστε μέσω των τροπολογιών του και ο εισηγητή. Αναφέρεται κυρίω στη δημιουργία και τη διατήρηση στην προστασία των θέσεων εργασία κάθε φορά που αναφερόμαστε στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Αυτά ουσιαστικά ήθελε να πει ο κύριο ε, Ντόιτ ή Γιούτα Στάνμπρουκ. Και πάλι εκ μέρου ε, τη που στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών ε, που λέει ότι ένας κρανισμός για την πρόσβαση τρίτων κρατών στις ε, κρατικές ε, συμβάσεις θα πρέπει να προβλέπει έναν διορθωτικό μηχανισμό που να επιτρέπει την αξιοποίηση ε, μέτρων κυρωτικών για εκείνα τα κράτη που προσπαθούν να ε, αξιοποιήσουν τι δυνατότητε μέσα στον στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρί αντίστοιχα να ανοίγουν, να ανοίγουν τι δικέ του αγορέ σε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με δικαιώματα και ελευθερίε των επιχειρήσεων, από ό,τι φαίνεται. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα που βρίσκεται η κοινωνική διάσταση, που βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Η κυρία Σίπλ καλωσορίζει την ε, γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότηση ε, του συναδέλφου κ. Ντόιτ ο οποίος ε, καταγράφει θέσεις πολύ σοσιαλδημοκρατικές, εντυπωσιακά σοσιαλδημοκρατικές, για σεβασμό των ε, συνθήκων, ε, συνθήκων εργασίας που άλλωστε έχουν ήδη θεσπιστεί μέσα από την οδηγία. Από την άλλη δεν βλάπτει να υπενθυμίσουμε κάποιες βασικές αρχές, γιατί για εμάς τους πάνω απ' όλα θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα θέματα της ε, απαγόρευσης της ε, πίεσης των ιδιωτικοποιήσεων. Θα πρέπει δηλαδή ο δημόσιος τομέας να αποφασίζει αν, ε, αυτόνομα αν σκοπεύει να προσφέρει μόνο του την υπηρεσία ή αν θα την εκχωρήσει. Η δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές θα πρέπει να ε, αφορά και τις περιπτώσεις της μαζικής παραβίασης των δικαιωμάτων εργαζομένων, όταν απαιτούνται κριτήρια αηφορίας, σεβασμό της ε, Σύμβασης του 1994, της Παγκοσμιονοχάρτης ε, Εργασίας και άλλες αντίστοιχες διατάξεις δεν πρέπει να επικρατούν μόνο μελήματα ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά θεμητού ανταγωνισμού Πρέπει να αποφύγουμε τις δυσμενείς για τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη διατάξεις και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των μειοδοτουσών προτάσεων πρέπει με έμφαση και προσοχή να επιβεβαιώνεται η τήρηση των ε, κοινωνικών εργασιακών συνθήκων. Η κυρία Σίπλη βρίσκει λοιπόν θετική την πρόταση γνωμοδότηση και προσβλέπει στην καλή συνεργασία με τον ε, συντάκτη και με τους λοιπούς και τους συγκητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο για τη συζήτηση. Όχι, από ό,τι βλέπω. Α, συγγνώμη κύριος Γκρόσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριος Κρότσμαν. Έχουμε το θέμα λοιπόν της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων για τις ε, δημόσιες ε, ε, αρχές. Δεν πρέπει να ανοίξει η αγορά κατά τρόπο ώστε να υπάρξει ανεξέλεκτη πρόσβαση, αλλά ούτε και προστατευτισμός. Χρειάζεται μια υγιής εμπορική πολιτική και με βάση το άρθρο 6 να βελτιωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ο κίνδυνος με νέα προστατευτικά μέτρα ε, να αντιδράσουν τα τρίτα κράτη όταν δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη έγκριση, να απέχουν δηλαδή ακόμη περισσότερο από την, αρχή της αμοιβαιότητας και υπάρχει κίνδυνο κίνδυνος της ε, του υγιούς ανταγωνισμού. Εάν, ε, εάν εγκρίνει τα μέτρα με βάση το άρθρο 10 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρίτα κράτη που παρεαβιάζουν τους κανόνες θα αποκλείονται από τις προκήρυξεις και τους διαγωνισμούς. Βεβαίως λοιπόν πρέπει να ενισχυθεί η θέση Επιτροπής στην υπόθεση αυτή, ε, αλλά με την προϋπόθεση της επιλογής ε, τις φθηνότερες λύσεις εφόσον αυτή δεν επιδεινώνει τις λοιπές συνθήκες. Οι διαδικασίες θα πρέπει να επιτρέπουν μια πρόσκοπτη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να θέτουν σε δυσμένες θέση τους Ευρωπαίους διαγωνιζομένους. Δεν πρέπει να ανατραπεί λοιπόν ο στόχος της ε, οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες που είναι η απλούστευση, η πιο διαφανής διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών και βεβαίως πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς μας υποχρεώσεις χωρίς να ε, η αγορά. εάν μία προσφορά δυνάμει του άρθρου 6 εξετάζεται, επαληθεύεται ε, ως προς την των προδιαγραφών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να οριστεί ένα εύλογο διάστημα και οι πληροφορίες σχετικές με την προ, ε, προέλευση πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα, αλλά όχι και κατά τρόπο που να αποκλείονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμό σε σχέση με επιχειρήσεις των τρίτων κρατών δεν είναι πρόβλημα. Είναι όμως πρόβλημα όταν είναι αθέμητος και μόνο τότε. Το υπογραμμίζω αυτό. Αθέμητο ανταγωνισμό όμως έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις όταν είναι παραδείγματι αποκλείονται ε, ορισμένες επιχειρήσεις ανεξαρτούς της προσφοράς τους. Υπάρχει δυνατότητα οι αθέμητες προτάσεις, η μη, ο μη θεμητός ανταγωνισμός να αποκλειστεί από τις διαδικασίες και αυτά τα μέσα που ήδη προβλέπονται πρέπει να αξιοποιηθούν. Θα πρέπει, όπως λέει και ο κύριος Ντότς, να αποκλείονται όσοι παραβιάζουν το ισχύον δίκαιο και Πρόκειται για διατάξεις οι οποίες ισχύουν και στο γενικό κανονισμό, δηλαδή οι φιλελεύθεροι είναι κατά των αθέμητων προτάσεων, κατά του dumping, αλλά όλα αυτά μπορούν να αριθμιστούν. Δεν δεχόμαστε λέει, τις προτάσεις όπως τις έχει περιλάβει η οδηγία. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρότσμαν. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Όχι. Ο κύριος Πίραστ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πώς θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τον πρωταρχικό στόχο της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί μερικές φορές ε, η πρόταση θεωρείται ως μέσο για να σταματήσουν οι συμβάσεις δημοσίων προμηθειών της Ένωσης. Αλλά αν εξετάσει εκ του σύνεγγυς τον κανονισμό αυτό, διαπιστώνει ότι το αντίθετο επιδιώκει. Γιατί εμεί θέλουμε το άνοιγμα των αγορών δημοσίων προμηθειών, των δημοσίων συμβάσεων. Και ιδιαίτερα αυτών που είναι κάτω των 5 εκατομμύριων ευρώ. Σε ό,τι αφορά τι δημόσιε συμβάσει που υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ώστε όταν απορρίπτεται μια προσφορά ε, θα πρέπει να οριθετούνται οι προϋποθέσεις για τέτοια απόρριψη. Τώρα, στις ε, δημόσιες συμβάσεις που είναι 7% των προμηθειών κάτω του κατοφλίου και εμπίπτωση στο πεδίο εφαρμογή οδηγίε, που είναι περίπου το 60% ε, της αξίας των συμβάσεων, δηλαδή από άποψη γραφειοκρατίας ακριβώς προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στις ε, πιο σημαντικές ε, συμβάσεις δημοσίων προμηθειών και με το άρθρο 6, τον αποκεντρωμένο μηχανισμό, δεν επιτρέπεται απόρριψη μιας προσφοράς ε, αν δεν εξεταστεί προηγουμένως η συνδρομή των προϋποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, μιλήσαμε για συγκεκριμένη επιφύλαξη σε περίπτωση δημόσ... Ε, διεθνούς συμφωνίας με εμπορικού εταίρου. Θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι τέτοιο εμπορικό εταίρο. Και επίση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχει σημαντική έλλειψη αμοιβαιότητας. Δηλαδή γίνεται ένας έλεγχος ουσιαστικά πραγματικός, ένας έλεγχος των πραγματικών συνθηκών που ξεπερνάει την απλή ύπαρξη ή έλλειψη τέτοιων διακριτικών, έλλειψη διακρίσεων και ελέγχουμε κατά πόσο οι συγκεκριμένες πρακτικές ε, οδηγούν σε διακρίσεις. Και αυτό το βρίσκουμε και στο άρθρο 6 για το επικεντρωμένο μηχανισμό και στο άρθρο 8 και, στα αρθρο 8 και 10. Θα πρέπει λοιπόν να ερμηνεύσουμε σωστά την πρόταση, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται και στο διατακτικό και, στην και στο αιτιολογικό της πρότασης. Επίσης, εξετάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή ε, τις προτάσεις σας για την ε, για ε, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η λήψη υπόψη κάποιων κοινωνικών ή περιβαλλοντικών κριτηρίων ήδη εξασφαλίζεται στα πλαίσια των βασικών οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες. Ενώ το συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη πρόταση δεν ε, ακυρώνει τους βασικούς κανόνες οι βασικές οδηγίες εφαρμόζονται και θα πρέπει να τηρούνται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Αλλά ο, ο κανονισμός, η πρόταση κανονισμού επικεντρώνεται στις προσφορές που γίνονται από τρίτες χώρες, από τελεστές τρίτων χωρών και που πληρούν τις προϋποθέσεις ή περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του κανονισμού. Υπό την επιφύλαξη φυσικά των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων που κατοχυρώνονται στις βασικές οδηγίες. Και που συζητούνται ακόμη στα πλαίσια της αναθεώρησης των ισχυσών οδηγιών. Είναι σημαντικά λοιπόν αυτά τα σημεία και θα πρέπει να τα έχετε υπόψη και στις μελλοντικές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητέ, να δώσω το λόγο στον κύριο Ρή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση γιατί φάνηκε μια αντιφατικότητα και μια διάσταση απόψεων. αλλά φαίνεται ότι παρόλο που ο εισηγητής προσπαθεί να σεβαστεί τη διάσταση απόψεων, ο ίδιος είναι καθόλου αντιφατικός, γιατί λαμβάνει υπόψη και τους ε, διεθνείς κανόνες που ισχύουν και για τις, δημόσι... για τις δημόσιες συμβάσεις και τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες και κριτήρια. Επίσης, τις συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού και το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων την ανάγκη αξιοπρεπούς εργασίες. Νομίζω ότι όλα αυτά τα σημεία ενισχύουν την κοινωνική διάσταση των βασικών οδηγιών και καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχόλια του εκπροσώπου των φιλελευθέρων, δεν είναι τυχαίο που στην εισαγωγή μου είπε ότι οι πιο ανοιχτέ δημόσιε συμβάσει του κόσμου είναι οι συμβάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση οι ανταγωνιστές μας, οι εμπορικοί μας ανταγωνιστές είναι πολύ προστατευτικοί στις αγορές τους. Οπότε εμείς προσπαθούμε να ανοίξουμε τις δικές μας αγορές προκειμένου να παρατηρούμε και τους εταίρους μας ε, να ανοίξουν τις δικές τους αγορές. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι ε, η προσέγγιση του εισηγητού μας είναι πολύ σωστή και εύστοχη. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής μας είναι πολύ συνεργάσιμος και περιμένει τις παρατηρήσεις ε, και τα σχόλιά σας. Και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί σας για την εκπόνηση κάποιων συμβαστικών τροπολογιών. Και φυσικά εμείς θα τις υποστηρίξουμε στην πολιτική μας ομάδα. Άσχετα με αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την λήψη υπόψη των κοινωνικών κριτηρίων και την ε, τη συμπερίληψη αυτών των δικαιών έμεσα στον κανονισμό των κριτήριων αυτών, θα πρέπει ο εισηγητή μα να εμβαθύνει στο σημείο αυτό και να το εξακριβώσει. Μέχρι τι 19 Απριλίου έχετε περιθώριο για να καταθέσετε τι τροπολογίε σα στι 12 το μεσημέρι. Η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου το Νοέμβριο θα εξετάσει αυτό το θέμα, οπότε έχουμε χρόνο. Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Τσάμπα Όρη για να μας παρουσιάσει την δεύτερη γνωμοδότηση του Thomas Deutsch με θέμα την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ή μάλλον την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, εξετάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος με θέμα την καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την βιοοικονομία στην Ευρώπη. Κύριε Ορίχη, το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, Στρατηγική Ευρώπη 2020 μάλλον. Και ξέρετε ότι η πράσινη οικονομία αποτελεί προτεραιότητα στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής. Είναι ένας τομέας όπου υπάρχει ένα δυναμικό ανάπτυξης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυναμικό ανάπτυξης όμως και για την απασχόληση και ιδιαίτερα θεωρούμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας χάρη στην λεγόμενη βίωη οικονομία. Γι' αυτό το λόγο ο συνάδελφος Deutsch θεωρεί ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο σημείο αυτό. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι φυσικοί πόροι όμως δεν αρκούν τελικά για όλους, δεν ανεξάντλητοι, Παράλληλα έχουμε και τις κλιματικές αλλαγές, οι οποίες πρέπει μακροπρόθεσμα να αντιμετωπιστούν. Όλοι αυτοί είναι πολύ διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν όμως το πρόβλημα αυτό. Πρέπει εμείς να βασιστούμε στην κοινοτομία, στην έρευνα, την επιστήμη και γι' αυτό το λόγο στο σχέδιο γνωμοδότησης ο Τάμας Ντόιτς εμένει στο ότι η βιοοικονομία μπορεί να συμβάλλει πολύ ευνοϊκά στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Δηλαδή μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή πλούτου, κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Η βιοοικονομία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ρήπανσης του περιβάλλοντος και μπορεί να συμβάλλει στο να δημιουργηθεί μία κοινωνία πιο ανταγωνιστική. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται επίσης στη γνωμοδότηση αυτή πάλι στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ο κύριος Ντόιτς αναφέρεται επίσης στην ε, ικανότητα καινοτομία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται μένα να θα πρέπει να ενδυναμωθεί, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να θέσει στην αγορά κάποια ανταγωνιστικά προϊόντα. Πρόκειται για μια σύντομη γνωμοδότηση. Και αναφέρθηκα απλώς στα σημαντικότερα αυτά σημεία τα οποία θέλει να τονίσει ο συντάκτη γνωμοδότη και προφανώ στη διάθεσή σα για περαιτέρω σχόλια. Ευχαριστούμε ο κύριος Στέρκας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ αντικαθιστώ την ε, συνάδελφο Αντιγόνη Παπαδοπούλου που προσπαθεί η κακόμερη να κατασβήσει την πυρκαγιά που προκάλεσε στην Κύπρο αυτή η υπεύθυνη ανεύθυνη που έχουμε στο Eurogroup. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας μεταφέρω την απόψη ε, της κυρίας Παπαδοπούλου. γνωμοδότηση του κυρίου Ντόμας Ντόιτς ε, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα και όλα όσα ακούσαμε από τον κύριο Τζαμπαόρη είναι σωστά και θα τα στηρίξουμε. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία που παραλείπονται και καλό θα ήταν να τα αναφέρουμε. Κυρίως δύο είναι αυτά που καλό θα είναι να αναφερθούν. Οι αλλαγές δεν θα πρέπει να γίνονται μόνο υπό το πρίσμα το ότι όλα είναι ρόδινα και τέλεια. Υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι και στις δύο πλευρές. Και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Γιατί έχουμε τεχνολογική επανάσταση και διαρθρωτικές αλλαγές που ανοίγουν νέους δρόμους και προοπτικές. Οπότε ε, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να προλάβουμε αυτές τις αλλαγές, όπως λέω και στη δική μου έκθεση για, για τις αναδιαρθρώσεις. Και επίσης ε, να φροντίσουμε να μην μείνουν κάποιοι εκτός νυμφών ή τουλάχιστον να μεριμνήσουμε για αυτούς. Και δεν θα πρέπει με το σύνθημα της βιοοικονομίας ή του πράσινων θέσεων εργασίας ε, και υπό, με το άλοθη της ε, ελαστικότητας να αγνοήσουμε στοιχειώδη σημεία της κοινωνικής νομοθεσίας. Καλή βέβαια η οικονομία, αλλά ακόμη και η οικονομία θα πρέπει να έχει κάποια κοινωνική πτυχή. Αυτή είναι η γνώμη των σοσιαλιστών. Οπότε θα συμπληρώσουμε την έκθεση του κ. Ντόιτς με κάποιες τροπολογίες για να περιλάβουμε πιο ισορροπημένα αυτό το νέο στοιχείο που ανακύπτει στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κύριος Βινιέ. Ναι, Πρόεδρε. Καταρχάς θα πρέπει να δηλώσω ίδιο συμφέρον ω ήθιστε τη σήμερα ημέρα, μια και ασχολούμαι με τη βιοοικονομία. Καλή είναι η έκθεση, γέννη. Κάποια στοιχεία θα θέλω να προσθέσω εγώ. Λεπτομέρειες για τη βιοενέργεια Στο σημείο 3 κατά πόσο πιθανότητα. Στο σημείο 7 για την ε, μαθητεία σε γενικέ εκμεταλλεύσει. Στην ύπεθρο καλύτερα για διάφορους, ε, ε, διάφορους τομείς ώστε να έχουμε ένα εργατικό δυναμικό κατερτισμένο καλά και με δεξιότητες που θα μπορούν να μεταφερθούν. Επίσης, το περιβαλλοντικό προϊόν πρέπει να εξετάζεται, όχι μόνο το εργασιακό για μια περιοχή. Πρέπει να κοιτάμε την ε, διατήρηση της βιοποικιλότητας που απαιτεί διάφορες δεξιότητες και ιδιαίτερα προς τη διαχείριση της ε, βιοπικιλότητας και ενισχύει τη βιοπικιλότητα. Αντί να οδηγεί σε απώλεια βιοπικιλότητας. Επομένως, στο σημείο 6 θα καταθέσω μια, μια τροπολογία. Αυτά έχω εντοπίσει προς το παρόν. Ίσως να βρω κι άλλα, βέβαια, δεδομένου ότι γνωρίζω τα πράγματα αρκετά καλά στον τομέα αυτό αν και θα προσπαθήσω να περιορίσω τις τροπολογίες μου σε ένα λογικό αριθμό. Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Η Επιτροπή. Παρακαλώ. Πολλό Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή Καλωσορίζω το ενδιαφέρον που εκδηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή μας. Καλώς ορίζει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης, διότι η απασχόληση διαδραματίζει κέριο ρόλο. Τα ζητήματα της γνωμοδότησης αποτελούν συστατικό τμήμα της διαδικασίας υλοποίησης στρατηγικής μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τις ε, απόψεις Επιτροπής ότι μπορούν να συμβάλλουν τα μέτρα αυτά στην δημιουργία ενώθου συνεργασία και την προαγωγή των ε, περιοχών της υπαίθρου με νέες δραστηριότητες ε, στηριζόμενες στις ανανεώσιμους πόρους, διαδικασίες νέες που μπορούν να αναζωογονήσουν ε, παράκτηση περιοχές της Υπέθρου και να δώσουν δυνατότητες όχι μόνο για τον Γιώργο και τον Αλιέα, αλλά και στη δευτεροβάθμια επεξεργασία, κατεργασία των προϊόντων, θέση εργασίας. Χρειάζονται βεβαίως δεξιότητες που μπορούν να απτυχθούν με συγκεκριμένα προγράμματα, με εκπαιδευτικά προγράμματα και είναι απαραίτητο η ε, ενημέρωση εχμής να είναι στη διάθεση του ε, ενδιαφερομένου για να κάνει λελογισμένες επιλογές. Το κοινωνικό πλεονέκτημα θα πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στις επιλογές της κοινωνίας και του χρήστη και ο καταναλωτής θα ενστερνιστεί την προστασία της βιοοικονομίας. Η στρατηγική μας στόχο έχει να εξασφαλίσει α, αλυσίδες ε, προμήθειας σε προϊόντα με σαφή παρουσία της βιοποικιλότητας Θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπορευσιμότητα των προϊόντων με μέτρα βελτίωσης ε, της πρόσβασης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με εφαρμογή της στρατηγικής βιοοικονομίας, τη βιοοικονομία 2020 και τη στρατηγική της, εν και του ορίζοντα 2020. Η δε δυνάμει επιτυχία της βιοοικονομίας στην Ευρώπη, θα βελτιώσει και την ανεξαρτησία μας από τα ε, ορυκτά καύσιμα, αλλά θα βελτιώσει και τις σχέσεις απασχολησιμότητας και γενικά τις οικονομικές συνθήκες για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ορή θέλει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που κάνανε όλες αυτές τις παρατηρήσεις οι οποίες θα διαβιβάσω στον κύριο Ντόιτσε. Από ό,τι βλέπω δεν νομίζω θα χρειαστεί να συζητήσουμε πάρα πολύ το όλο ζήτημα. Η συνεργασία είναι ήδη πάρα πολύ καλή και πολύ επικοδομητική. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταφέρουμε πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε το κείμενο αυτό και ελπίζω ότι το τελικό κείμενο θα σας βρει όλους σύμφωνους. Πάντως θα διαβιβάσω στον κύριο Ντόιτς όλες τις σημερινές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη, ο κύριος Μπά κανονικά είναι ο εισηγητής και μου είπε ότι έρχεται κυρία Πρόεδρε, φτάνει σε λίγα λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε να διοργανώσω καλύτερα τη συνεδρίαση. Πάντως, για την έκθεση του κυρίου Ντάτσε πρέπει να σας πω ότι ε, η το 26 Μαρτίου 5 το απόγευμα είναι η ημερομηνία κατάθεσης των τροπολογιών και το Μάιο θα ψηφίσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπακ, ο οποίος μόλις έφτασε και μας επιτρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να εξετάσουμε και το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο θα συζητήσουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή για την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Πρόκειται για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Αρμόδια καθήλυνη επιτροπή είναι η Επιτροπή Μεταφορών και εισηγητή στην Επιτροπή αυτή είναι ο κύριος Μαρινέσκου. Κύριε Μπακ, λοιπόν, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι έφτασα πραγματικά τελευταία στιγμή. Θα μιλήσω γερμανικά. Όπως έχω συνηθίσει. Έχουμε να κάνουμε ένα σημαντικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δυναμικό που δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη. 5,1 εκατομμύριο είναι η θέση εργασίας, 2,4% επί του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ συγκεκριμένα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα απολογισμό μετά τον απολογισμό του 2005 όπου προβλέπει προόδους ε, στις αερομεταφορές σημειώνει σημαντικές προόδους χωρίς όμως επιτρέψη των στόχων. Οχτώ χρόνια μετά την το τελευταίο απολογισμό και μετά την νέα κρίση, το κλίμα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Η κρίση έχει ε, επηρεάσει σημαντικά το χώρο των αμερομεταφορών, έχει προβάλλει νέες προέγαλες προκλήσεις για την αγορά. Η Ε, ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές αερομεταφορών βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, ενώ εμπόδια στην εσωτερική αγορά παραμένουν, εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αποδιαρθρωθούν για να λειτουργήσει απροσκοπτά η εσωτερική αγορά. Υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες νομικές, ε, φορολογικές και άλλες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρόκειται για εμπόδια στην εσωτερική αγορά, πρόκειται για συνθήκες οι οποίες ε, μπορούν να επηρεάσουν και τον, ε, το επίπεδο επιβάρυνση των αεροδρομίων, την ασφάλεια, γενικά την ανταγωνιστικότητα των αερομεταφορών της Ευρώπης. Και μας ως Επιτροπή Απασχόλησης ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει να διαφυλαχθούν υψηλέ προδιαγραφές εργασία. Στι συμφωνίε, λοιπόν και με τρίτες χώρες πρέπει αυτέ οι αξίε προδιαγραφές και βέλτιστες πρακτικές ή περιβαλλοντικέ προδιαγραφές να τηρούνται, να γίνονται Χωρίς τόσο και η απελευθέρωση να οδηγήσει στην ε, υποβάθμιση των υψηλών προδιαγραφών εργασίας ή προσχέσεις του περιβάλλοντος. Εδώ έχουμε να κάνουμε φυσικά με μια πολύ λεπτή ακροβασία, ένα σπαγκάτο θα έλεγα. Γιατί και έτσι πρέπει να υποστηρίξουμε τον ε, ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό και να μεριμνήσουμε ότι δεν αποβαίνει αυτό εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των προδιαγραφών εργασίας. Ξέρετε ότι έχω ένα περιθώριο, ένα όριο 1500 χαρακτήρων για τη γνωμοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν θα με ευγνώμων σε οποιοδήποτε συνάδελφο θέλει να βελτιώσει το κείμενο χάρη σε νέε τροπολογίε. 27 του μηνό, προθεσμία για τροπολογιών. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μπένιον Στάινμπρουκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τα σχόλιά του. Συμφωνώ με αυτά που άκουσα μέχρι στιγμής. Αυτή τη φορά την πρόσβαση στην αγορά και την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς, πολύ σημαντικά θέματα, ενιαίοι ευρωπαϊκοί εθέρες, επίσης σημαντικό θέμα, γιατί έτσι γίνεται ανταγωνιστικός ολόκληρος ο κλάδος και προς τα έξω. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν θα πρέπει να γίνει μία κούρσα προς τα κάτω σε ό,τι αφορά τους ε, κανόνες ε, για την απασχόληση. Μια ευθύνωσα πορεία δηλαδή. Δεν θεωρώ όμως ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο εφόσον ε, εφαρμοστεί σωστά η ισχύουσα νομοθεσία και αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε. Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, σίγουρα χρειάζεται καλή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και μια τέτοια νομοθετική μεταρρύθμιση ήταν ευπρόσδεκτη. Ίσως όμως το σχετικό σημείο παρά είναι φιλόδοξο και θα προσπαθήσω να το μετριάσω με τις τροπολογίες μου. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τις θετικές πλευρές της κατάστασης και το πιθανό δυναμικό σε θέσεις εργασίας. Να, να συνδέσουμε τους κόμβους με την χώρα δημιουργώντας έτσι πιο ανταγωνιστική οικονομία και θέσεις απασχόλησης. και στο εσωτερικό αλλά και σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και να δημιουργήσουμε δελεστικές όρους και προϋποθέσεις και για να προσελκύσουμε επιχειρήσεις και για να όχι μόνο για να εγκατασταθούν σε εμάς αλλά και για να παραμείνουν. Γι' αυτό και θέλουμε σωστή διασύνδεση των αεροδρομίων των αστικών κέντρων, των σημαντικών κόμμων με την Εδοχώρα. Γιατί η Εδοχώρα για να γίνει ελκυστική για τις πολυεθνικές εταιρείε και για εσωτερικές επενδύσεις θα πρέπει να είναι καλά να εξυπηρετείται δεόντως και από αεροπορικές γραμμές. Και θα καταθέσω και τέτοιες τροπολογίες. Η κυρία Στάιμπουκ. Ναι, ευχαριστώ. Ακούσαμε τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσίασε ο Σόξμπαχ. Και βέβαια αυτά αποδεικνύουν από μόνο του πόσο μεγάλη σημασία έχει ο χώρο, ο τομέα των αερομεταφορών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είτε πρόκειται για, την, ε, για τα σχόλια τα φορολογικά, είτε πρόκειται για την δημιουργία και ασφάλεια ή εξασφάλιση τη εργασία. Ε, εάν δούμε βέβαια και τα θέματα που μας απασχολούν εδώ στην Επιτροπή τα θέματα που θα θέλαμε να εξετάσουμε στην Επιτροπή εργασία, είτε πρόκειται για τα αεροδρόμια, είτε πρόκειται για τι Υπηρεσίε Εδάφου, τι ώρε εργασίας των πιλότων και του, προσωπικού, του πληρώματος ε, του προσωπικού ε, θαλάμου Καμπίνα ε, που έχουμε δει πρόσφατα. Βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συνθήκες εργασίας και πόσο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον ε, πολύ διεθνή ανταγωνισμό διαφυλάσσοντας και τις θέσεις εργασίας, τις ε, ε, εταιρείε αεροπορικές, τα αεροδρόμια και αυτό με ε, συμφωνίες για την πολιτική των αεροματοφορών. Γιατί εάν δεν μεριμνήσουμε εγκαίρως κινδυνεύουμε να χάσουμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας ε, απελήθησαν, ε, χάθηκαν το 2012 μόνο από το χώρο των αερομεταφορών ε, από τις ευρωπαϊκές εταιρείες εκτός Ευρώπης. Ο αυτό που μας λέει ουσιαστικά είναι ότι δεν μπορούν όποιες ρυθμίσεις συμφωνίες να συνάπτονται εις βάρος των εργαζομένων. Αυτό το θεωρούμε ευπρόσδεκτο. Επρόσδεκτη είναι λοιπόν η γνωμοδότηση του κυρίου Μπαχ και ιδιαίτερα καθώς υπογραμμίζει τι κοινωνικές πτυχέ, τι παραγράφου 4, 5 και 6, το πρόβλημα που έχουμε είναι ο στρεβλός ανταγωνισμός στον χώρο των αερομεταφορών, στη σχέση ευρωπαϊκή Ένωση με τα τρίτα κράτη τη Ασία, τη ε, Μέση Ανατολή, τη Άπου Ανατολή και την ε, δυνατότητα για προαγωγή μιας κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των αερομεταφορών. Πολύ σημαντικό είναι, και χαίρομαι που και ο Παχ δεν το παραμέλησε, είναι το θέμα των χαμηλών αμοιβών στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πρέπει να οδηγήσει σε, μια, σε έναν αγώνα δρόμο προς τα κάτω, σε μια συνεχή μείωση των αμοιβών. Ξέρουμε ότι και η Αραβική Χερσόνησος είναι μια από τις περιοχές που ε, ανταγωνίζεται ε, τις δικές μας αεροπορικές εταιρείες αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επικρατήσουν συνθήκες που δεν είναι βιώσιμες για τον Ευρωπαίο εργαζόμενο. Η αεροπορική εταιρεία και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τηρεί τις, τα βασικά δικαιώματα, δικαιώματα του συνεταιρίζεις, του συνέρχεστε, την αναγνώριση των συλλογικών συμβάσεων, τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής ε, και όλες αυτές τις συνθήκες που έχει επιβάλει η σχετική σύμβαση του οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Πρέπει να ισχύουν λοιπόν αυτές τις συνθήκες και πιστεύω ότι όλοι είμαστε πλέον επαρκώς ευαισθητοποιημένοι ώστε και να γνωρίζουμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις εταιρείε μας, αλλά και ταυτόχρονα καθήκον της Επιτροπής μας είναι να προστατέψει πάνω απ' όλα τον εργαζόμενο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει το λόγο. Ουδής, λοιπόν, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε ηγητά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αερομεταφορών είναι μια υπηρεσία, ένας κλάδος μάλλον που δημιουργεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει ουσιαστικά να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για τους δικούς μας αερομεταφορείς, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κοινοτικό επίπεδο γίνεται στα πλαίσια του ενιαίου ουρανού, αλλά ξέρετε ότι σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν και διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Όσον αφορά κυρίως αυτή την εξωτερική πτυχή, η ευρωπαϊκή πολιτική για τις αερομεταφορές επικεντρώνεται σε κάποιες συμφωνίες όπου θα πρέπει να υπάρχουν ρήτρες κατά της διακρατικής μεταχείρισης, ιδίως όσον αφορά την ε, πρόσβαση σε κάποια τέλη αεροδρομίου ή όσον αφορά τις χρονοθυρίδες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να ισχύουν τα ίδια κριτήρια με αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος, για τον ισότιμο ανταγωνισμό, για την προστασία του καταναλωτή και έχουμε επίσης και την ε, οδηγία εφαρμογής των ε, ευρωπαϊκών, ε, μάλλον την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον χρόνο εργασία. η οδηγία αυτή η κοινοτική θα ισχύει και συμφωνίε οι οποίε συνάπτουμε με τι όμορφε μα χώρε. Επίσης, κατά την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων που έχουμε, προσπαθούμε να εμπλέξουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από τον κλάδο και εφόσον το δέχονται οι χώρες εταίροι μπορούν και αυτές να συμμετέχουν ως παρατηρητές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ που στην έκθεσή σας ε, αναφέρεστε στο ότι αρχίζει να αναθεωρείται ο κανονισμός 868 του 2004 όσον αφορά την προστασία των ευρωπαϊκών εταιριών από, τους, από τις αθέμητες συνθήκες ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μελετήσει τις διάφορες εναλλακτικέ που υπάρχουν προκειμένου να καταλήξει σε ένα πιο αποτελεσματικό μέσο και να προστατεύσει κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερο τις ευρωπαϊκές εταιρείε σε σχέση με τον αθέμητο ανταγωνισμό ή την ευνοϊκρατία που μπορεί να έχουμε σε κάποιες άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε σχέση με του εθνικού αερομεταφορεί των χωρών αυτών θα είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό προκειμένου να επιβάλλουμε τα ίδια κοινωνικά πρότυπα και στις άλλες χώρες. Πάντως ε, βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της όλης διαδικασίας και θα προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε όλο και περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εκπόνηση αυτού του νέου κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θέλει να υπάρχει και μια συγκεκριμένη ρήτρα θεμητού ανταγωνισμού η οποία να συμπεριλαμβάνεται στις διμερείς συμφωνίες οι οποίες συνάπτουν τα κράτη-μέλη με χώρες εταίρους. Πέρα από όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση κατά την προετοιμασία και το συντονισμό της ευρωπαϊκής κοινή θέσης κατά την διάσκεψη την οποία διοργανώνει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας αναφερθήκαμε στον ισότιμο ανταγωνισμό και η Ιρλανδική Προεδρία ανέλαβε πραγματικά να προωθήσει τη θέση αυτή, λέγοντα ότι θέλουμε σε όλε τι διμερεί συμφωνίε να έχουμε αυτή τη ρήτρα ισότιμου ανταγωνισμού, στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Euh, euh, Κύριε Μπαχ, θέλετε να ξαναλάβετε το λόγο. Δεν έχω πολλά να προσθέσω νομίζω. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους, τις συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως για την παρουσίαση τις παρατηρήσεις, τις ε, πληροφορίες μας έδωσε για περαιτέρω προτάσεις. Θέλουν να εμπλέξουν και τους κοινωνικούς εταίρους και βέβαια το κοινοβούλιο και χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία. λαμπρά. 20 Μαρτίου το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες, μια και η Επιτροπή Μεταφορών θα αποφαθεί το Μάιο. Οπότε θα έχουμε στο μεταξύ των χρόνων να εγκρίνουμε και εμείς τη δική μας γνωμοδότηση. Εξαντλήσαμε την απόγευμα την ημασημέρι σε διάταξη. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και βράδυ και σας δίνω ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί και μην ξεχάσετε τις κάρτες ψηφοφορίας.